Colleagues, if I can open Ξεκινάμε τη συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη καταρχήν του. Σας ευχαριστώ. Μετά έχουμε τα πρακτικά της 30 Σεπτεμβρίου και της 14 Οκτωβρίου. Και αν δεν έχετε αντίληψη, τα εγκρίνουμε όλα αυτά. Ανακοινώσεις Προέδρου. Καμία ανακοίνωση δεν έχω να σας κάνω. Διορισμοί εισηγητών και σκιωδών και συντακτών ε, γνωμοδότης θα τα πούμε αυτά αύριο μετά τις συνεδρίες των συντονιστών το βράδυ. Περνάμε τώρα στα εναλλακτικά καύσιμα, την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων. Η εξέταση των τροπολογιών έχει έρθει ο κύριος Φιντάντσα ή ακόμα. Θα περιμένουμε μια στιγμή να έρθει ο κύριος Φιντάντσα. Ήρθε ο κύριος Φιντάντσα. Πάολο, περνάμε στην εκθεσή σου για την ανάπτυξη εναλλακτικών ε, καυσίμων. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Το θέμα αυτής της έκθεσης είναι το ακόλουθο. Είχαμε 317 τροπολογίες από τους συναδέλφους, αρκετά σημαντικό αποτέλεσμα που δείχνει έντονο ενδιαφέρον για το θέμα. Ανέλησα αυτές τις τροπολογίες ε, μία-μία. Πολλές από αυτές τις θεωρώ θετικές και ευθυγραμμεζόμενες προς τις ε, δικές μου παρατηρήσεις. Ε, πάνω στο έργο αυτών των τροπολογιών έχω εμπιστοσύνη, νιώθω σίγουρος ότι θα συζητήσουμε μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία έτσι ώστε να προχωρήσει αυτός ο φάκελος από μέρους του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ φιλόδοξο και ρεαλιστικό το εγχείρημα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κινούμαστε σε ένα πλαίσιο έντονου σκεπτικισμού σε πολλά κρατη Δεν είναι απλές οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Επί της ουσίας, ορισμένα σχόλια, αναθέμα, σύμφωνα με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Ένας αριθμός τροπολογιών αφορά τις ημερομηνίες για την επίτευξη των στόχων. Πάνω σε αυτό, στο σχέδιο έκθεσης, δεν έχω λάβει συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή, δεν τροποποίησα τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ασφαλώς αυτό θα είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που θα πρέπει να συζητήσουμε με τους σκιώδεις εισηγητές ε, στο πλαίσιο και των ε, διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να έχει ένα περιθώριο ελιγμών. Μια άλλη ομάδα τροπολογιών αφορά τα εθνικά στρατηγικά σχέδια συμφωνώ με πολλές από αυτές, ιδίως εκείνες που προβλέπουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να αναπτύξουν εθνικά σχέδια με διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εναλλακτικά καύσιμα και εγγυόμενα μια τεχνολογική ουδετερότητα, χωρίς να ξεχνούμε ότι η αγορά αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την άποψη της έρευνας και της τεχνολογίας. Θα πρέπει φυσικά να λαμβάνουμε υπόψη τον αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει να εγγυηθούμε μια στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών, μελών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και του κλάδου. Και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών σχεδίων. Όσο αφορά τις τροπολογίες ε, για την ηλεκτρική ε, ενέργεια, πολλοί συνάδελφοι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη εγγύησης, εξασφάλισης των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα, στην αγορά όπως έχει σήμερα. Ε, θεωρώ ότι πρόκειται για έναν κατανοητό στόχο παρόλο που θεωρώ ότι δεν πρέπει να χάνουμε από τα μάτια μας τον βασικό μας στόχο, ο οποίος είναι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να έχουμε μια ενοποιημένη ομοιόμορφη κατάσταση που θα επιτρέπει στους χρήστες των κρατών μελών να χαίρουν των ίδιων προδιαγραφών στο δίκτυο σε όλες τις χώρες. Για τους στόχους τώρα, Πιστεύω πως πρέπει να έχουμε υποχρεωτικούς στόχους. Ασφαλώς θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και ίσως πιο ρεαλιστικοί με βάση το κείμενο της Επιτροπής. Ε, σίγουρα λοιπόν μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ μιας κάποιας ευελιξίας, μεγαλύτερης ευελιξίας διατηρώντας ε, τη γενική αρχιτεκτονική της πρότασης. Υπάρχουν συγκεκριμένες τροπολογίες, για παράδειγμα για τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στα αεροδρόμια, ε, όταν ε, τα αεροπλάνα βρίσκονται σε κατάσταση στάθμευσης, όταν παραμένουν ακίνητα στην πίστα. Ως προς το δεύτερο παράρτημα, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες κάποιοι συνάδελφοι ε, ζητούν απάλληψη του παραρτήματος, όλου του παραρτήματος. Αυτό σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να το δω με τους σκιώδεις εισηγητές. Γιατί εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν συγκεκριμένοι στόχοι και υποχρεωτικοί στόχοι. Ε, η αφετηρία μου λοιπόν ε, μάλλον καταρχήν είμαι κατά της απάλληψης του παραρτήματος και είμαι κατά το να γίνουν οι στόχοι προαιρετικοί. Θεωρώ ότι οι υποχρεωτικοί στόχοι αποτελούν βασικό κομμάτι του προγράμματος αυτού. Όσο αφορά το υδρογόνο, υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες ε, που εκφράζουν νομίζω μια αλφα μηχανία απέναντι στο, στο εφικτό χρήσης αυτής της τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα. Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Μετά υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο αέριο, το υγραέριο. Ε, νομίζω ευθυγραμμίζονται με το πνεύμα της έκθεσής μου οι τροπολογίες αυτές. Οπότε ασφαλώς θα μπορέσω να τις εντάξω σε αρκετά αντιπροσωπευτικούς συμβιβασμούς με τους διαφόρους συναδέλφους. Υπάρχουν και άλλα συγκεκριμένα θέματα που θα μπορούσα να αναφέρω. Το άρθρο 7, το θέμα της ενημέρωσης προς τους καταναλωτές. Όλοι συμμεριζόμαστε την ανάγκη να, να υπάρχουν διαφανείς και σαφείς πληροφορίες προς τους ε, καταναλωτές ως προς τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων και γι' αυτό θα ήθελα πολύ να μπορέσω να υπάρξουν και άλλα μέτρα υπέρ των καταναλωτών. Υπάρχει και ένα θέμα παρόμοιο ε, για το παράρτημα 3, όπως το θέμα που τίθεται για το παράρτημα 2, όσο αφορά τις προδιαγραφές, τα πρότυπα, και πάνω στο θέμα αυτό νομίζω προς την ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Αντίθετα, υπάρχει ένα μέρος που αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού για την ε, μεταφορά επικίνδυνων φορτίων στους εσωτερικούς πλωτούς δρόμους. Εκεί υπάρχει ένα στοιχείο αγοράς. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου στις, στα εσωτερικά πλωτά ύδατα, ε, στα, στις εσωτερικές υδάτινες μεταφορές. Και θα δούμε κατά πόσο αυτή η πρόταση αναθεώρησης πηγαίνει προς την ευκταία κατεύθυνση, δηλαδή την κατεύθυνση της εγγύησης μιας μεγαλύτερης δυνατότητας χρήσης αυτής της μορφής φυσικού αερίου για να λυθεί και το πρόβλημα αυτό της μεταφοράς του στα εσωτερικά ύδατα. Αυτά είχα να πω για τις προτάσεις ε, για τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Όπως είπα θα συναντηθώ με τους ε, σκιώδεις εισηγητές και θα προσπαθήσω να καταλήξω σε συμβιβαστικές προτάσεις. Πάνω στα ειδικότερα θέματα τώρα θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή και με το γραφείο του καθενός για να δούμε αν θα μπορέσω να ετοιμάσω κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Μα ικανοποιεί σε γενικέ γραμμέ η πρόταση του εισηγητή. Μόνο μερικέ ε, προσθήκες θα θέλαμε να κάνουμε υπομορφή τροπολογιών. Καταρχήν αυτά τα οποία μπορούμε να υποστηρίξουμε απόλυτα. Η ενίσχυση η οποία πρέπει να γίνει στον εθνικό χώρο στρατηγική για τα θέματα αυτά για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στο σημείο αυτό, να υπάρξουν ενδιάμεση στόχοι και σε εθνικό επίπεδο και ιδίω να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω πλήρω τη θέση του εισηγητή στα σημεία αυτά. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο πιστεύω θα, θα χρειαστεί περισσότερη προσοχή σε ό,τι αφορά τα εθνικά υποδείγματα για την ηλεκτροκίνηση που θέλουμε να υποστηρίξουμε, αλλά εκεί θα πρέπει να μας ενδιαφέρει από ποιες πηγές παράγεται ο ηλεκτρισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για την ε, ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή θέλουμε να μην παράγονται από πυρηνική ενέργεια ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιείται, αλλά από πράσινες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν και ποιες είναι οι επιπτώσεις που θα προέλθουν από την δημιουργία αυτής της νομοθεσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα βενσινάδικα τα οποία είναι οικογενειακά ή είναι μικρές επιχειρήσεις και τα οποία δεν πρέπει να υποστούν ιδιαίτερη πίεση από αυτή την οδηγία επιπλέον. Εγώ θέλω να χαιρετήσω το γεγονό ότι ο κ. Φιντάλτσα υποστηρίζει το να υπάρχουν δεσμευτικοί και ποσοτικοί στόχοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το υποστηρίζω. Πρέπει πράγματι να είναι δυνατόν να έχουμε μια υποδομή η οποία θα επιτύχει αυτούς τους ποσοτικοποιημένους και δεσμευτικούς στόχους. Κάτι άλλο όμως το οποίο θέλω να εξετάσει ο εισηγητής και όπου πρέπει να βρούμε κάποια λύση όλοι, είναι να έχουμε διατυπώσεις οι οποίες δεν θα αποδυναμώσουν την ε, διαφάνεια και την δεσμευτικότητα όταν λέμε λοιπόν για ενδεικτικού στόχου ή για στόχου, στο περίπου, όλα αυτά για μένα αποτελούν αποδυνάμωση και επομένω δεν νομίζω ότι αυτά μπορούν να συμβάλλουν σε μια μεγαλύτερη ασφάλεια σε ό,τι αφορά τι επενδύσει στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν και εμεί από νομική άποψη να, μην έχουμε σαφείς διατυπώσει να μην περάσουμε σε μια φαιά ζώνη και να μην αποδυναμώσουμε την πρόταση. Αυτό το οποίο θα ήθελα να υπάρχει σαν συμβαστική πρόταση είναι σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, έχει προτείνει να υπάρχουν ε, ποσοτικοποιημένοι στόχοι για το 2020, 2020. Θέλει να φτάσουμε το 5% στα ηλεκτρικά αυτοκείμενα σε ό,τι αφορά τις νέες ταξινομήσεις σε κάθε κράτος μέλος μέχρι το 2020. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό, αλλά θέλω να εξασφαλίσω ότι αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος είναι ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος. Να διατηρήσουμε λοιπόν αυτό το στόχο, αλλά να θεωρήσουμε σαν ε, δεδομένο το, σαν κατώτατο επίπεδο το 3% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι 5% γιατί υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες στα κράτη-μέλη. Είναι πολύ διαφορετική η αγοραστική δύναμη στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη όπου είναι περιορισμένη η αγοραστική δύναμη των πολιτών να υποχρεώσουμε τους πολίτες να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία γενικά είναι πολύ δάπανα. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό και γι' αυτό το λόγο εγώ θα ήθελα να κατεβάσω το 5% προτείνει Κομισιόν σε 3% ποσοστό ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα αυτό είναι το πιο σωστό και ένα ακόμα σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω για την υποδομή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε για το πώς θα συνδεθεί αυτό με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δηλαδή, στους ε, λιμένες οι οποίοι συνδέονται με τα διευρωπαϊκά δίκτυα να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν υποδομές <clears throat> για να υπάρξουν και δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Γιατί αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, πάλι καταλήγουμε σε μια αμφίσιμη αντιμετώπιση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και δεν συνάδει κάτι τέτοιο με αυτά τα οποία έχουμε προτείνει μέχρι τώρα. Αυτά είναι λοιπόν οι προτάσεις μου και εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένο και ζητώ και την υποστήριξη όλων να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε οι ποσοτικοί στόχοι που βρίσκονται στη Λευκή Βίβλο για το διοξείδιο του άνθρακο θα μπορέσουν να πάρουν δεσμευτικό χαρακτήρα και να μπορέσουν να συμπεριληφθούν και στις κατευθυντήριες γραμμέ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Για μένα είναι λοιπόν πολύ θετικό ότι ο ΣΥΤΙΣ προωθεί την εναρμόνιση των ε, πριζών τύπου 2 για την ηλεκτροκίνηση και εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει και μια έγκριση από την Επιτροπή Τυποποίησης. Να υποστηριχθεί λοιπόν αυτή η, η λύση και φυσικά η λύση θα πρέπει να είναι διαλειτουργική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Εκεί που τώρα διαφέρω λιγάκι από τον εισηγητή είναι η έννοια των ελαχίστων <clears throat> ε, υποδομών για το LPG, για το υγροποιημένο προπάνιο, για το υγραέριο. Αυτό δεν είναι ένα πράσινο ε, καύσιμο, είναι ένα παραπροϊόν της διήλυσης του πετρελαίου και επομένως είναι ένα ορυκτό καύσιμο. Δεν πρέπει εμεί να υποστηρίξουμε λοιπόν την χρήση του υγραερίου αυτού σαν πράσινου καυσίμου. Κατά τα άλλα όμως συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία ζητάει ο εισηγητής. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Όταν αρχίσαμε τη συζήτηση, είχαμε πέντε ομιλητέ, τώρα πήγαμε στου εννέα. Δέκα αυτή τη στιγμή. Έχουμε 30 λεπτά για το συζήτηση του θέματο. Το είχαμε ξανασυζητήσει. Δεν θα φτάσει η ώρα. Οπότε, αν μπορείτε να είστε συνοπτικοί στι παρατηρήσει σα και σύντομοι. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί νομίζω ότι η έκθεση αυτή έχει πολλά ικανοποιητικά στοιχεία. Μίλησα και για το θέμα αυτό την προηγούμενη φορά. Εγώ έχω καταθέσει 10 τροπολογίες και άλλοι το έχουν πράξει. Σε γενικέ γραμμέ, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον συγητή. Έχει δίκιο ο κύριο Φιντάντσα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την τεχνολογική ουδετερότητα για τα θέματα αυτά. Αυτό είναι απαραίτητο σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση που θέλουμε όλοι να την προωθήσουμε αλλά φυσικά, όπω είπε και ο κ. Σέρτου, έχει σημασία από πού έρχεται η ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να προέρχεται από ηλεκτρικέ, από ε, συγγνώμη, ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας και επίσης είναι σημαντικό να έχουμε και μια εναρμόνιση για τις πρίζες τύπου 2. Αλλιώς είναι μια βλακία να μην έχουμε καμία ε, διαλειτουργικότητα. Δεν πρέπει να ρισκάρουμε να μην έχουμε αυτή τη διαλειτουργικότητα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να σκεφτούμε και τη χρήση της ηλεκτροκίνησης στα αεροδρόμια για να μειωθεί και ο θόρυβος ο οποίος δημιουργείται. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία κινούνται στα, στην πίστα των αεροδρομίων να μπορούν να κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και μπορούμε απλώς να το υποστηρίξουμε πλήρως. Για τις ελάχιστες τώρα απαιτήσει για το ε, υγραέριο, και εγώ αντιμετωπίζω τα ίδια προβλήματα με τον κύριο Ερτού και το είπα και την προηγούμενη φορά, δεν πρόκειται για ένα εναλλακτικό καύσιμο το LPG, το υγραέριο. Ξέρω ότι μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, αλλά δεν είναι εναλλακτικό καύσιμο και έχουμε ήδη μια υποδομή για το, για το καύσιμο αυτό. Και εδώ πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί για το πώ θα πάρουμε θέση σε σχέση με τι τροπολογίε για το υγροποιημένο. Τώρα φυσικό αέριο, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στους λιμένε υπάρχει η απαραίτητη υποδομή και αυτό ισχύει και για τους λιμένε εσωτερικών ε, υδατίνων δρόμων και φυσικά πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και για τα φορτηγά να μπορούν να μεταφέρουν αυτό το φυσικό αέριο. Νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ και προσβλέπω στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για τα περαιτέρω. Κύριο Στέιλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Δεν δυσκολεύομαι να συμφωνήσω με τον κύριο Φιντάντζα ότι θα μπορούσαμε να τυποποιήσουμε τα συστήματα διασύνδεσης και παροχής. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δούμε και τι στόχους υποκρύπτουν αυτές οι επιλογές και οι υποδομές για τα εναλλακτικά καύσιμα. Νομίζω ένας στόχος είναι αυτό που αναφέρει και η Λευκή Βίβλο, να μειωθούν οι εκπομπέ διεξιδίου του άνθρακα από τι μεταφορέ κατά 60% στο 2050. Κατά την άποψή μου, το πώ θα φτάσουμε αυτό το στόχο από τη σημερινή κατάσταση, αυτό που προτείνεται δηλαδή να επιδιώξουμε χρησιμοποιώντας τις υποδομές για τα εναλλακτικά καύσιμα, δεν αποδεικνύεται για την ώρα, δεν είναι σαφές ότι αν ακολουθήσουμε την οδό που προτείνει ο κ. Φιντάντσα θα καταλήξουμε όντως να πετύχουμε μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση όμως. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και επίσης βλέποντας τι γίνεται με τα εναλλακτικά καύσιμα, να σκεφτούμε και το πώς θα πρέπει να αλλάξει η χρήση των μεταφορών. Να περάσουμε από τα ε, κλασικά μεταφορικά μέσα στα λεωφορεία, τα τραμ, τα τρένα, τα ποδήλατα και το περπάτημα. Το θέμα όμως είναι να αναρωτηθούμε, θα πετύχουμε κάτι με όλα αυτά. Αυτό που λέμε εδώ είναι πώς θα, να, αυτό που προτείνεται εδώ είναι πώς θα δαπανηθούν για τα εναλλακτικά καύσιμα και τις υποδομές τους πολύ μεγάλα δημόσια κονδύλια, κρατικά κονδύλια, χωρίς να ξέρουμε στο τέλος τι θα πετύχουμε. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζήτηση, την υπερβολική ζήτηση. Και δεν το ξέρουμε, διότι η αγορά, πούμε, για τα ηλεκτρικά, για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί. Ή δεν ξέρουμε τι ακριβώ θα γίνει με τη χρήση ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια ή ενέργεια ηλεκτρικής ενέργειας η ενεργεια που προερχεται απο τις ανανεώσιμες πηγές. Ε, η παροχή ε, φυσικού αερίου λόγω χάρη τα σημεία ανεφοδιασμού σε βενζίνη. Θα πρέπει να επενδύσουμε δημόσια χρήμα ή τέλος πάντων επιτρέψουμε να επενδύσει δημόσιο χρήμα σε κάτι που είναι τόσο αμφίβολο αποτελέσματος. Και επίσης να επιστήσω την προσοχή σας σε μια μεγάλη εταιρεία ιαπωνική λιανική, εταιρεία ελληνικής πώληση που έχει επενδύσει σε σημεία ανεφοδιασμού ε, σε όλη την Ιαπωνία. Για φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Η έκθεση εδώ ζητά κάτι ανάλογο από το Κοινοβούλιο. Εγώ θα έλεγα να αφήσουμε την, ε, τους ιδιώτες, τη βιομηχανία να κάνει αυτές τις επενδύσεις. Όμως θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ο στόχος μείωσης εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα ε, μπορεί να ε, επιτευχθεί καλύτερα με την επένδυση δημόσιου χρήματος σε αυτές τις υποδομές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μπορούμε να στηρίξουμε τον εισηγητή. ιδίω για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ένα δίκτυο που ελπίζουμε ότι θα επεκταθεί και γι' αυτό δεν υποβάλαμε και σχετικέ τοπολογίε. Νομίζουμε ότι στο σχέδιο τη έκθεση αναφέρεται πολύ σωστά. Επίση, ένα-δυο σημεία τα οποία ήθελα να σχολιάσω. Η δεσμευτικό χαρακτήρα των σημείων φόρτιση ευαίσθητο θέμα. Ε, εδώ νομίζουμε ότι πάμε πολύ μακριά και γι' αυτό έχουμε υποβάλλει την τροπολογία 125 που ζητά να επιτευχθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ των υψηλών φιλοδοξιών μας και του ρεαλισμού όμως που θα πρέπει να έχουμε στην προσέγγιση μας. Ελπίζουμε να το λάβει υπόψη ο εισηγητής. Επίσης όλη η συζήτηση για, τους, ε, ε, για τη διασύνδεση και το κατά πόσον μπορεί να αξιοποιηθούν η έκθεση θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις που όμως να φανούν ε, επιτυχημένες και, στη, και για την αγορά. Και έτσι θα καθοριστεί το κατά πόσον ε, μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή όχι. Ε, θα ήθελα να ζητήσω και από εσά και από τον εισηγητή να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην 246. Αυτό για τα σημεία TNT Μιλάμε για τα σημεία ανεφοδιασμού και φόρτιση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τροπολογία 246, πιστεύω. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Πιστεύω ότι η οδηγία για τις την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μα από ορυκτά καύσιμα. Φυσικά πρέπει να έχουμε και εναλλακτικά σχέδια δράση για τα εναλλακτικά καύσιμα προ το παρόν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε του στόχου αυτού που έχουμε θεσπίσει. Γι' αυτό θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε ορισμένε από τι τροπολογίε που εγώ υπέβαλα. Κατέθεσα μια τροπολογία καταρχήν για να υπάρχει η έννοια του σταθμού επαναφόρτισης. Δηλαδή να υπάρχουν σταθμοί φόρτισης που έχουν στον πληθυντικό, που είναι πολύ ε, που έχουν πολλά σημεία φόρτισης, να μπορεί επομένως να επαναφορτίζεται παραπάνω από ένα αυτοκίνητο κάθε φορά. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να επαναφορτίζεται γρήγορα, άλλο να επαναφορτίζεται με πιο αργό ρυθμό και κατέθεσε επίσης και τροπολογίες που αφορούν τις νέες ε, <clears throat> προδιαγραφές που θα αφορούν τα σημεία επαναφόρτησης για τα νέα αυτοκίνητα. Στην Εστονία, για παράδειγμα, έχουμε ένα σχέδιο προς την κατεύθυνση αυτή. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο επαναφόρτησης το οποίο να καλύπτει όλη μας τη χώρα. Δεν θέλουμε να πάνε χαμένες οι επενδύσεις για αυτό το δίκτυο και έχω καταθέσει επίσης και τροπολογίες για τον αριθμό και την πυκνότητα των σημείων επαναφόρτης. Η κυρία Φώστρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και πολλές ευχαριστίες στον εισηγητή για τη σκληρή του δουλειά. Δυστυχώς ε, δεν συμφωνούμε με αρκετά πράγματα, ε, με αρκετές τροπολογίες, αλλά δεν συμφωνούμε κατά ανάγκη και με τις ε, παραδοχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκονται πίσω από αυτήν την έκθεση. Ε, η γενική μας θέση στις αρχικές μας συζητήσεις ήταν ότι ό,τι και αν θα συμφωνούσαμε στο τέλος θα έπρεπε να κατευθύνεται από την αγορά. Ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να κάνει αυτό που επιθυμεί και βέβαια η ευθύνη του κράτους μέλους είναι να στήσει την υποδομή που θα το επιτρέψει αυτό. Γενικά λοιπόν το 2020 είναι πολύ πρόωρη χρονική στιγμή για την ε, ανάπτυξη αυτής της υποδομής. Ωστόσο θεωρούμε ότι είναι καλό να υπάρχει, να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνεται η συζήτηση γιατί προχωράει και ο κόσμος της τεχνολογίας. Ε, έχω σημειώσει μερικά πράγματα, ορισμένες τροπολογίες. Την 376. Η Επιτροπή φαίνεται ότι πιστεύει πως ε, οι μπρίζες τύπου 2, οι γερμανικές, αυτές, ότι αυτές πρέπει να προωθήσουμε, ενώ αναφέρθηκε ήδη το παράδειγμα της Ιαπωνίας και επίσης το σύστημα που χρησιμοποιεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην Μάνχη αυτή τη στιγμή. Ελπίζω λοιπόν η Κομισιόν να μην θελήσει να επιβάλλει ένα και μόνο προϊόν. Θα πρέπει η αγορά να μπορεί να επιλέξει αυτό που θέλει, όποια, τεχνολογία θέλει. Η 205, η ανάπτυξη της υποδομής μέχρι το 2020, αυτό το ανέφερα βέβαια. Και πάλι, ε, δεν είμαστε βέβαιοι για τον αριθμό των ηλεκτρικών ε, αυτοκινήτων, οπότε είναι πρόωρο σε κάθε περίπτωση να το συζητούμε από τώρα. Τέλος, ε, ο εισηγητής είναι υπέρ των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Εμείς είμαστε κατά. Θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν τα ίδια τις πολιτικές τους και τον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων και υπάρχουν και τα θέματα της επικουρικότητας και της γεωγραφίας και πρέπει να διατηρήσουμε μία ευελιξία. Εξετάζουμε και συνυπολογίζουμε και τη θέση της αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος. Ε, δεν το λέει ρητός πουθενά η έκθεση, αλλά επειδή μιλούμε για δισεκατομμύρια, αν όχι τρισεκατομμύρια ε, ευρώ, τότε θεωρούμε, ότι, θεωρούμε πως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάντως θα πρέπει να συνεχίσουμε την συζήτηση οπωσδήποτε, αλλά είναι πολύ πρόωρο να επεκτείνουμε αυτές τις υποδομές αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει για την έκδοση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Φιντάντσα. Κύριε Σκόμε. Μα και εμείς υποστηρίζουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και έχουμε φιλόδοξους στόχους για τις μεταφορές 20% μείωση έναντι του 1990 να κάνουμε εξοικονόμηση σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος έναντι του 2000, το 2020 έναντι του 1990. Γιατί βλέπουμε ότι στον τομέα των μεταφορών έχουν αυξηθεί οι εκπομπές αντίθετα με τη βιομηχανία. Αλλά δεν λύνουμε το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Με την... Η κίνηση με τα οχήματα έχει πέντε ε, μειονεκτήματα, η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος που μπορεί να λυθεί με την ηλεκτροκίνηση, αλλά αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλη την αλυσίδα από την παραγωγή της ενέργειας μέχρι την χρήση της. Και αυτό δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Τα αυτοκίνητα τα παραδοσιακά μειώνουν κατά 25%, μπορεί να μειώσουν κατά 25% τις εκπομπές τους, εάν χρησιμοποιήσουμε καλύτερα υλικά για, την, για τον κίνδυνο, για τον ε, θόρυβο. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο αθόρυβα σε, χαμηλό, σε χαμηλή ταχύτητα, αλλά σε υψηλή ταχύτητα είναι το ίδιο. Το κόστος τώρα του δικτύου. Ουσιαστικά εμείς ε, επιδοτούμε κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 1.600 ευρώ. Δεν μπορούν να πλησιάσουν τις τιμές των συμβατικών αυτοκινήτων δεν θα αλλάξει η χρήση των αυτοκινήτων των ηλεκτρικών. Τίποτα στα θέματα των ατυχημάτων και η, γερμανική, η ομοσπονδιακή ε, Γερμανία έχει αποφασίσει να μειώσει το, την κάλυψη από δρόμους και από άσφαλτο σαν ποσοστό του εδάφους της ε, επικράτειάς της. Οπότε ούτε και με αυτόν τον τρόπο δεν λύνουμε το πρόβλημα. Φυσικά το φυσικό αέριο είναι καλύτερα από την βενζίνη ή το πετρέλαιο, αλλά ακόμα και το φυσικό αέριο ουσιαστικά κάποτε θα εξαντληθεί. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μας κάνουν σκεφτούμε διαφορετικά, να σταματήσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Καλές είναι οι ανανεώσιμες ενέργειες, αλλά 20% της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος προέρχονται από την αποψήλωση του τροπικού δάσους. Εγώ βλέπω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αποτρέψουμε με την πορεία που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, αλλά να έχουμε μια συνολική εικόνα για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει λοιπόν να δίνουμε επιδοτήσεις κρατικές για τα θέματα αυτά. Με, πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει η οικονομία της αγοράς να αντιμετωπίσει. Γιατί πρέπει τώρα να παίρνει τόσα λεφτά η αυτοκινητοβιομηχανία για να προωθήσει την ηλεκτροκίνηση. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι πολύ παλιά η ηλεκτροκινητικότητα το 1881 ξεκίνησαν οι πρώτοι ηλεκτρικοί, τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ στο Βερολίνο. Δεν είναι καινούρια ιδέα, δεν μπορεί κανείς να το παρουσιάζει μετά από 130 χρόνια σαν μια κοινοτομία την ηλεκτροκίνηση. Και είναι απαραίτητη η ουδετερότητα σε σχέση με την χρήση των τεχνολογιών. Αλλά εγώ τονίζω ότι αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ε, κινητικότητα, δεν θα προστατεύσουμε το κλίμα του πλανήτη μας. Και εδώ κλείνω. Πρέπει να σκεφτούμε ένα διαφορετικό τρόπο άλλες τεχνολογίες για τα αυτοκίνητα. Για τα λεωφορεία, για τα μικρά φορτηγά. Αν είναι καλύτερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εντάξει. Και γι' αυτό πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα για τις πρίζες και τους υποδοχείς σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να γίνει και για τα πλοία. δεν μπορεί λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα αυτό της ρήπανσης παρά μόνο αν εφαρμοστεί και στα πλοία στον βαθμό του δυνατού αυτή η αντιμετώπιση. Ο κύριος Δεγκράντες, σας ευχαριστώ. Οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Κομισιόν από την πρότασή της, που την υποστηρίζει ο εισηγητής, Εγώ θα εξηγήσω τώρα ποια είναι η θέση μου σε σχέση με όλα αυτά. Νομίζω ότι σε μια εποχή οικονομικής κρίσης θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές το να δημιουργήσουμε νέες πολυδάπανες υποδομές αυτή τη στιγμή δεν είναι η πιο λογική λύση. Επιπλέον, αυτές οι υποδομές θα οδηγήσουν σε πάγιο κόστος. Είναι απαραίτητο να είμαστε πιο επιφυλακτικοί όταν εμείς σχεδιάσουμε νέες υποδομές για τα ενεργειακά αυτά ζητήματα. Και επιπλέον, πιστεύω ότι ο ρεαλισμός αυτός θα είναι πολυθετικός και αυτά θα τα δούμε με τον συγητή. Θα αναφερθώ τώρα στι τροπολογίε μα. Έχουμε προτείνει μερικέ τροπολογίε, οι οποίες διαφοροποιούν τη θέση μας εναντί του εισηγητή. Υπάρχουν δυσκολίες στην εμπορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γι' αυτό έχουμε ζητήσει ο αριθμό των ε, σταθμών επαναφόρτηση να τροποποιείται κάθε χρόνο σε σχέση με τον αριθμό των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν και τι προβλέψει για περαιτέρω πώληση. Δεύτερον, θεωρούμε ότι η επαναφόρτιση θα πρέπει να γίνεται με χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει και ευφυής χρήση σταθμών επαναφόρτισης και ιδιωτικών χώρων ε, ε, επαναφόρτησης. Μια καλύτερη χρήση λοιπόν της τεχνολογία. Και έχουμε προτείνει και μια τροπολογία σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι σταθμοί επαναφόρτησης. Και ο συγητής έχει παρουσιάσει κάτι αντίστοιχο, επομένως νομίζω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση για τους σταθμούς φυσικού, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είπαμε ότι αυτή η σταθμή δεν πρέπει να είναι κατά ανάγκη ε, σταθερή και για την επαναφόρτιση σε υδρογόνο. Η Κομισιόν λέει να υπάρχει ε, το 2020 παντού ένα σταθμό επαναφόρτιση μέσα σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων. Εμείς θέλουμε τα κράτη-μέλη επί τη βάση της αίτησης για χρήση υδρογόνου να μπορούν να εξασφαλίσουν το 2030 την πλήρη κυκλοφορία των οχημάτων με υδρογόνο στο έδαφος. Αυτά. Κυρία Σαναλόβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Συγκεκριτή για τη δουλειά του. Είναι πολλά τα σημεία μετά που μπορούμε να συμφωνήσουμε, όμως θέλω και εγώ να κάνω κάποια σχόλια για τρεις τροπολογίες. Μία από αυτές τάσεται υπέρ των στόχων προσανατολισμού περισσότερο στόχων ενδεικτικών και όχι δεσμευτικών για τα σημεία φόρτισης αυτό το 2020. Το 10% των σημείων αυτών ε, προτείνεται να είναι κρατικά. Η δημιουργία όμω ε, των υποδομών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τι τοπικέ ανάγκε, τι τοπικέ αγορέ, καθώ και το τι είδου χρήστε υπάρχουν. Αυτό στις τροπολογίε 216 και 223. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας εδώ στην τροπολογία 237 η οποία αφορά τους τελικούς χρήστες που ήδη έχουν αγοράσει ηλεκτροκίνητο όχημα βάσει των σημερινών ε, προτύπων επαναφόρτησης. Αυτοί θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα κατά τη ε, διάρκεια κύκλου ζωής του οχήματός τους να μπορούν να χρησιμοποιούν το ισχύον σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Τροπολογίε για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έχω αποβάλει και εγώ ε, και αυτέ θέλω να σχολιάσω. Νομίζω πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα εγχώρια σημεία φόρτιση θα είναι τα βασικά για τα ηλεκτροκινητά οχήματα. Οπότε, ναι, συμφωνώ, χρειάζονται στόχοι, αλλά θα πρέπει να είναι και λογικοί. Δεν θέλουμε να δαπανίσουμε υπερβολικά πολλά κονδύλια για υπέρμετρο αριθμό σημείων φόρτιση. Άλλωστε, πρέπει να σκεφτούμε ότι οι απαιτήσει για κρατικά σημεία φόρτιση δεν θα είναι ίδιε όπω για ιδιωτικά σημεία ή τέλο πάντων ε, σημεία που έχουν δημιουργηθεί με ιδιωτικό χρήμα, ιδιωτικέ επενδύσει. Για την τροπολογία του εισηγητή, την τροπολογία 44, για την ευθύ μέτρηση ή την απομάκρυνση τη ευθύου μέτρηση. Μου λένε από την Ήτρα ότι αυτό ίσως να αντιφάσκει με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι στην Ήτρα έχουν βρει μια συμβαστική λύση για το άρθρο 4,6 για την ευθύ μέτρηση. Ελπίζω ο εισηγητής να βρει χρόνο να το δει και αυτό διότι είναι τελευταία στιγμή ε, πρόταση και μπορεί να μην είναι συμβατό με την νομοθεσία, όπως προτείνεται. Για την λειτουργικότητα νομίζω είναι καθοριστική σημασία στο σημείο αυτό και όπως είπε η κυρία Φώστερ, Έχουμε τουλάχιστον δύο διαφορετικά μοντέλα που λειτουργούν ταυτόχρονα στην Ευρώπη και νομίζω ότι θα είναι σημαντικό για τα κρατικά σημεία φορτισής, τα δημόσια σημεία φορτισής, να προτείνονται και τα δύο μοντέλα, τα δύο πρότυπα. Είναι πολύ, εύκολα, πολύ εύκολο με τα τεχνολογικά μας μέσα να χαρτογραφήσουμε το που βρίσκονται τα διάφορα σημεία. Αν το παρακάνουμε όμως θα έχουμε πολλά αυτοκίνητα που δεν θα μπορούν να κουνηθούν και να μετακινηθούν στην Ευρώπη. Δεν έχει λοιπόν νόημα να υπερβάλλουμε στην δημιουργία σημείων φόρτισης. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται αν προταθούν νέα τεχνολογικά σημεία μέσα μάλλον που θα απαιτούν την προσαρμογή των σημείων φόρτισης που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Οπότε να είμαστε αρκετά ευέλικτοι. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Μπένιον. Εγώ ίδιος να πω σύντομα ότι ενώ συνήθως ε, συμφωνώ με τον κύριο Κράμερ, δεν ε, έχω και μονή με τα ηλεκτροκινητά οχήματα που θα πρέπει να είναι το μελλοντικό κατεξοχήν μέσο ιδιωτικών μεταφορών. Υπάρχουν και τα θέματα των ε, σημείων φόρτισης και το θέμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για το συνδρομικό δίκτυο λέγαμε πάντοτε ότι είναι το πιο περιβαλλοντικά φιλικό μέσο μεταφοράς γιατί είναι ηλεκτροκίνητα τα τρένα, αλλά τους πυρηνικούς σταθμούς, ας πούμε, ή τα εργοστάσια άνθρακα. Τι θα τα κάνουμε. Οπότε στο μέλλον πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα γιοταχή ε, και αν θα είναι όλα ηλεκτροκίνητα. Δεν λέω να μην υπάρχουν εναλλακτικέ. Σίγουρα θέλουμε εναλλακτικέ για τα ορυκτά καύσιμα, αλλά κάτι που με ανησυχεί, α πούμε, είναι, ω προ την έκθεση αυτή, ότι φαίνεται να οδεύουμε προ τον ηλεκτρισμό. Είναι καλή η ηλεκτρική ενέργεια για να οδηγούμε και ε, τα εναλλακτικά καύσιμα, μάλλον το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είναι μόνο εναλλακτική για του λιμένε. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Διότι εάν δείτε τι γίνεται με το μεθάνιο, υπάρχει ένα 25% επένδυση εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να το αξιοποιεί. Γιατί δεν αρέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μεθανόλη. Για τις θαλάσσιες μεταφορές υπάρχει εδώ μετατροπή κατά 25% της μεθανόλης. Ε, εμείς δεν το αναφέρουμε καν. Περίεργο δεν είναι. Και επίσης για το γαλποποιημένο φυσικό αέριο. Η αποθήκευση του φυσικού αερίου, του υγροποιημένου, πώς θα το αποθηκεύουμε. Σε κάποια τραγικά χαμηλή θερμοκρασία πρέπει να ε, αποθηκεύεται. Πώς θα την πετυχαίνουμε αυτή την τόσο χαμηλή θερμοκρασία, σε τι είδους περιέκτη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί μην τα πετάξουμε όλα εδώ στο ίδιο καλάθι, ε, μακροπρόθεσμα να έχουμε ως στόχο μόνο την ηλεκτρική ενέργεια και να είναι η μόνη μας επιλογή για τις οδικές μεταφορές και για τις θαλάσσιες μόνο το ευρωπημένο φυσικό αέριο. Ας μας πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η μεθανόλη δεν αναφέρεται λόγου χάρη. Μία εναλλακτική πηγή ενέργειας θέλουμε ή πολλές για τις ανάγκες των μεταφορών μας. Πέραν αυτού, βεβαίως όλοι συμφωνούμε να μειωθούν οι εκπομπές. Βεβαίως όλοι θέλουμε να απαγκιστρωθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Αλλά να επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Κράμερ. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα απομονωμένα, λες και το υπόλοιπο σκηνικό ή το οποίο δεν ισχύει. Ολόκληρη την αλυσίδα ανεφοδιασμού πρέπει να, λέμε, να βλέπουμε πριν πούμε ότι το τάδε μέσο είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον ή το περισσότερο καθαρό και ούτω καθεξής. Κύριε Ονίλη. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατανοείτε ότι από τη δική μου οπτική το γεγονός ότι η λίστα των αγορητών πήγε από τους 5 στους 10 είναι πολύ θετικό. Καταρχήν ευχαριστώ. Ε, σχόλια του Προέδρου Εκτός μικροφώνου. Ναι, πάνω από 10 αγορητές, πράγματι. Δεύτερον, ε, βλέπουμε ότι προκαλέσαμε ενδιαφέρον όχι μόνο από τον αριθμό των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί, αλλά βλέπουμε και την εξαιρετική ποιότητα των τροπολογιών και μπορώ να πω ευθύς εξ αρχής ότι με ελάχιστες τροπολογίες θα διαφωνούσαμε. Και αυτό είναι μια ειλικρινής ε, ένδειξη ε, της εξαιρετικής δουλειάς που έχει γίνει πάνω στην πρότασή μας. Θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της πρότασής μας. Η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης ε, βελτιώνει πάρα πολύ την ε, πρότασή μας. Ε, στα περισσότερα σημεία υπάρχει σύμπνια. αρκεί να υπάρξουν πέντε τμήματα πέντε όψεις. Χρειαζόμαστε δεσμευτικά εθνικά πλαίσια. Κυρία Φώστερ, δεν είπα ευρωπαϊκά ενοποιημένα ομοιόμορφα πλαίσια, εθνικά πλαίσια. Ε, πράγματι γίνεται μια απόπειρα ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς, αλλά με βάση τις εθνικές, οι οποίες καθοδηγούνται από κάποια κοινά στοιχεία. Θέλουμε να ενισχύεται και όχι να υπονομεύεται η εσωτερική αγορά, η ενιαία αγορά. Ε, λοιπόν, ε, μάλλον υπάρχει περιθώριο ανάλογα με το πόσο αυστηροί είμαστε ως προς τους στόχους. Όμως τους στόχους τους χρειαζόμαστε. Ορισμένοι το θίξατε το θέμα αυτό. Δεν πρόκειται να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις εάν δεν υπάρχει κάποιος βαθμός προβλεψιμότητας ε, η οποία να εκφράζεται σαφώς στα εθνικά στρατηγικά σχέδια σε βάθος κάποιων ετών. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το έτος 2020 είναι η σωστή οπτική, η σωστή προοπτική από την πλευρά των χαρακτών πολιτικής σίγουρα θα πρέπει οι αριθμητικοί στόχοι που προτείνονται, να, οι ποσοτικοί στόχοι που προτείνονται να βελτιωθούν ή να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Για τους σταθμούς επαναφόρτισης ε, ε, μπορούμε να επικεντρωθούμε ε, στα δημόσια σημεία επαναφόρτισης και να μην ασχοληθούμε με τα ιδιωτικά σημεία επαναφόρτισης. Επίσης, Πρόεδρε, ε, θα θέλαμε να διασφαλίσουμε όλες τις εναλλακτικές ε, προτάσεις και καύσιμα. Η μεθανόλη. Δεν έχουμε τίποτε κατά της μεθανόλης. Απλώς ε, κατά το χρόνο που προετοιμάζαμε την νομοθεσία αυτή. Δεν είδαμε να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο, στο συγκεκριμένο καύσιμο, στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Νομίζω όμως ότι το σχέδιο έκθεσης πραγματικά εκφράζει μια διάθεση να συμπεριληφθούν όλα τα εναλλακτικά καύσιμα και όλες οι κατηγορίες μεταφορών. Ε, τρίτον, χρειαζόμαστε πρότυπα και προδιαγραφές, ενιαία πρότυπα και προδιαγραφές, διαφορετικά δεν θα υπάρξει ενιαία εσωτερική αγορά και τα αναλλακτικά καύσιμα. Τούτου λεχθέντος, ασφαλώς είμαστε πολύ ανοιχτοί ως προς το μεταβατικό στάδιο για τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη κάνει πολλές επενδύσεις σε διαφορετικό πρότυπο η προδιαγραφή. Ας πάρω το παράδειγμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός ότι προτείνεται να υπάρξει ένα ενιαίο πρότυπο ε, κατά τρόπο που έστω ε, να αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα να έχουμε σταθμούς επαναφόρτισης ε, με δύο πρότυπα ταυτόχρονα είναι κάτι που μπορούμε να το δεχτούμε. Αρκεί στο τέλος της διαδικασίας να κινηθούμε όλοι προς ένα ενιαίο πρότυπο. Αυτό είναι ζωτικό νομίζω. Ε, επίσης, για τους καταναλωτές, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνουν κάποια ουσιώδη μέτρα για τους καταναλωτές. Όλοι έχουμε δει τις δυσκολίες με την ένταξη των βιοκαυσίμων, όπου οι καταναλωτές ε, ε, περιέπεσαν σε πλήρη σύγχυση, δεν ήξεραν αν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για τα οχήματά τους κτλ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κάποια απλά μέτρα, ε, σαν αυτά που προτείνουμε εμείς, αλλά και ο εισηγητής και η Επιτροπή σας. Τώρα, για τον χρόνο. Ε, παρακαλώ, ας μην Ας μην πάμε μέχρι το 2030. Θεωρούμε ότι μία σειρά βασικών επιλογών πρέπει να γίνουν μέχρι το 2020. Ε, κάποιες από τις υποχρεώσεις, για παράδειγμα για το υγροποιημένο αέριο, στις θαλάσσιες μεταφορές, ίσως θα μπορούσαμε, ε, όπως προτείνατε μερικοί, ε, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τα για το πλέγμα των διευρωπαϊκών δικτύων, γιατί εν τέλει αυτός, είναι ο κόμβος τον οποίο προσπαθούμε να χτίσουμε. Το 2020 λοιπόν είναι απολύτως ουσιώδες και να έχουμε και κατά νου ε, ότι ορισμένες από τις δεσμεύσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές και πάλι οι τρεις ε, ζώνες θείου, όχι μόνο στη Βαλτική, αλλά και στη Μεσόγειο, ε, για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις εδώ και τώρα και όχι με την προοπτική του 2030. Τέλος, μια από τις ε, πρόσθετες ιδέες που ήρθαν στο προσκήνιο με τις τροπολογίες, να μην υπάρξει πρόσθετο οικονομικό βάρος για τους ε, κρατικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Ε, είναι ορθό να γίνει αυτό επί της αρχής και υπήρξε και σημαντικό κομμάτι των συζητήσεων. Εμείς προσπαθούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό και να το συνυπολογίσουμε όταν αποφασίζουμε για τους ποσοτικούς στόχους, γιατί αυτό είναι ουσιώδες και για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Από την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι είναι καλή πρακτική να τονίσουμε το γεγονός ότι στην έκθεση αυτή δεν απαιτούνται πρόσθετη εθνική πόροι. Σας ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Φιντάντζα, ευχαριστώ. Ο πλούτος της, ε, του διαλόγου που είχαμε με καθησυχάζει και μάλιστα πολύ περισσότερο από τον προηγούμενο γύρο συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους που ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικές. Είναι πολλά τα θέματα που γέρθηκαν και Νομίζω με τους κοιόδης εισηγητές θα καταφέρουμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Βεβαίω δεν είμαι αφελής. Δεν πιστεύω ότι με αυτή την οδηγία θα λύσουμε ε, το πρόβλημά μας διαπαντός ή αυτομάτως θα πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει στην περιβαλλοντική μας πολιτική μέχρι το 2050. Και εγώ είμαι ρεαλιστής στην προσέγγισή μου και αντιλαμβάνομαι ότι μόνο εν μέρη αυτή η παρέμβαση με αυτή την οδηγία θα πετύχει κάποια αποτελέσματα. Όμως, συνολικά και σε σχέση με μια σταθερή αγορά αυτή των ε, εναλλακτικών καυσίμων, υπάρχει ανάγκη να υπάρξει και ένα συγκεκριμένο σημείο αφετηρίας. Ιδάλλως, θα έχουμε διαρκώς το δίλημα και το ερώτημα του αυγού και της κότας. Δηλαδή, υποδομές ενώ δεν υπάρχει αγορά ή η αγορά δεν υπάρχει γιατί δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές. Νομίζω το να έχουμε θετική στάση όπως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το να ξεκινήσουμε από ένα συγκεκριμένο σημείο αφετηρίας. Δηλαδή να εντοπίσουμε την ανάγκη ενός σταθερού νομοθετικού πλαισίου για να επιτρέψουμε και να μπορέσουν να γίνουν οι κατάλληλε επενδύσει είτε κρατικέ και δημόσίε με κοινοτικά εργαλεία ενδεχομένω, εφόσον χρειαστούν συγκεκριμένε ε, υποδομέ για τα ενελεκτρικά κάψιμο, όπως είπε ο κ. Χέρτουκ, για το ε, προγραμματισμό TNT ω προ τα ε, θέματα αυτά και για την δημιουργία υποδομών ώστε παραλληλώς να μπορέσει να αναπτυχθεί και η σχετική αγορά. Νομίζω λοιπόν από αυτήν την έννοια θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Για αυτά που είπε ο συνάδελφος Τέιλορ. Το αν είμαστε βέβαιοι ότι οι προβλέψεις αυτές μπορούν να έχουν και συγκεκριμένο αντίκτυπο αριθμητικό στην μείωση των εκπομπών του διοξιδίου. Αυτήν τη βεβαιότητα δεν μπορώ να σας την δώσω εγώ. Όμως, ε, παρακολουθώντας την εξέλιξη της πρότασης οδηγίας, είχαμε και μια μελέτη... Ε, μελέτη σκοπιμότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε κατά πόσο οι προβλέψει αυτέ είναι ρεαλιστικέ ή όχι. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για το θέμα των λιμένων και τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η θέση μου διαφέρει λίγο από αυτή κάποιων συναδέλφων. Θεωρώ ότι από τη μηδενική ανάπτυξη των υποδομών αυτή τη στιγμή μέχρι το να προβλεφθεί υποχρεωτικά να υπάρχουν σημεία ανεφοδιασμού ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου σε όλους τους λιμένες ε, της σχετικής συμφωνίας νομίζω είναι σημαντικό. Βέβαια πρέπει να υπάρξει και ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Εγώ έρχομαι από μια χώρα όπου οι λιμένες ε, καλύπτονται από τη συμφωνία τέντη. Χρειάζεται όμως και μεγαλύτερη κρατική συμμετοχή για την ε, ανάπτυξη αυτών των λιμένων. Δεν μπορούμε να αφήσουμε όλη την ευθύνη στα κράτη-μέλη για να καλύψουν τις ανάγκες των λιμένων. Νομίζω λοιπόν από αυτή την άποψη δεν θα πρέπει να προβλέψουμε υπερβολικά άχθη για τα κράτη-μέλη. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, διότι με απειλείτε με το σφυράκι σας. Για ορισμένα ζητήματα νομίζω θα διαφωτιστούμε περισσότερο μετά τη συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές, αλλά σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση όλους για την συμμετοχή σας και τις συνεισφορές σας. Ευχαριστώ. 26 Νοεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία. Εάν ο εισηγητής μπορεί να συνεννοηθεί με τους σκιώδεις και να καταλήξουμε σε συμβασικές τροπολογίες, μπορεί να καθυστερήσει, αλλά καταρχήν λέμε 26 Νοεμβρίου για την ψηφοφορία. Ως προβλεπόμενη ημερομηνία σας ευχαριστώ όλους. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα. Αγορά μεταφορής πακέτων, παράδοσης πακέτων για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 20 λεπτά έχουμε καθυστερήσει. Παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Κύριε Νταντέν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω ότι η έκθεση αυτή υπογραμμίζει τις οικονομικές επιπτώσεις από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τονίζει τρία σημεία που υπάρχουν ελλείψεις, η έλλειψη διαλειτουργικότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών και έλλειψη πληροφόρησης προς τον καταναλωτή. Κατατέθηκαν 55 τροπολογίες, επί τη βάση των οποίων εγώ μπορώ να σας προτείνω 6 συμβιβαστικές τροπολογίες που καλύπτουν 39 από τις 55 αυτές τροπολογίες. Οι τροπολογίες αφορούν την παράγραφο που έχει να κάνει με την πληροφόρηση των καταναλωτών, την καλύτερη διαλειτουργικότητα και την καλύτερη λειτουργία των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα του ανταγωνισμού για τα ταχυδρομεία, την ανάπτυξη των ετικετών και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών. Οι περισσότερε πολιτικέ ομάδε έχουν συμφωνήσει για τι συμβαστικέ αυτέ τροπολογίε. Εγώ δεν Έχω παρά μόνο λίγε τροπολογίε για τι οποίε εγώ προτείνω αρνητική ψήφο, γιατί νομίζω ότι απομακρύνονται από το στόχο τη Επιτροπή μα και μου φαίνεται ότι προχωρούν πάρα πολύ ε, προ μία κατεύθυνση ή προ την άλλη. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σύντομο. Ευχαριστώ κύριε Ντάντεν. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπατε και πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάισνα. Και εγώ πάρα πολύ σύντομα μπορώ να τα πω. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του και τον κύριο Φιντάντσα ήθελα να ευχαριστήσω, αλλά έφυγε προηγουμένως. Πράγματι, σε πάρα πολλά σημεία συμφωνούμε ιδιαίτερα <clears throat> και εμείς δεν έχουμε καταθέσει πάρα πολλές τροπολογίες. Αυτά τα οποία ζήτησα νομίζω ότι έχουν καλυφθεί από τις συμβαστικές τροπολογίες. Είναι εύστοχε λοιπόν οι συμβαστικέ τροπολογίε και μπορώ να πω ότι έχει κάνει πολύ καλή εργασία ο εισηγητή στη γνωμοδότηση αυτή και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Περιμένουμε την ψηφοφορία. Κυρία Λίχτεμπέργκερ, και εγώ συμφωνώ με το μεγαλύτερο μέρος των συμβαστικών τροπολογιών του κυρίου Νταντέν. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλά. Μόνο μία αίτηση, αν θέλετε, έχω να κάνω. Στην ε, συμβαστική τροπολογία D είχα αναφέρει εκεί ότι όλα αυτά τα οποία θα αποφασιστούν εδώ δεν πρέπει να στρέφονται κατά τις στοχοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος. Γιατί εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, κίνητρα για την παράδοση πακέτων σε, μικρό, σε μικρότερες παρτίδες κτλ. Γι' αυτό έχω προσθέσει μια πρόταση που λέει ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε σύγκρουση με τους υφιστάμενους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των, ε, της, κίνησης φορτίων σε, και την επιβάση του περιβάλλοντος επειδή θα μετακινούνται πάρα πολύ μικρά, για πάρα πολύ μικρά φορτία πακέτα. Κύριο Στάιν από την ε, Γενική Διεύθυνση Αγοράς. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νταντάν. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για μια πάρα πολύ καλή και ισορροπημένη έκθεση η οποία πραγματικά ευθυγραμμίζεται με όσα έχω δει, με όσα έχω ακούσει. Εξακολουθούμε να δουλεύουμε πάνω στην πρωτοβουλία παρακολούθησης ε, σε συνέχεια όσων έγιναν το περασμένο έτος, αλλά μπορώ να σας πω ότι από τη μία πλευρά δεν πρόκειται να προτείνουμε καινούρια νομοθεσία η οποία να αναστατώσει τις αγορές σε αυτή τη χρονική στιγμή. Από την άλλη πλευρά ακούμε με ευαισθησία ε, όλα όλες τις προτάσεις που έχουν να κάνουν με την αηφορία. Αν διαβάσετε την πράσινη βίβλο θα δείτε ότι εξ αρχής τα είχαμε εντάξει όλα αυτά. Ε, Ποτέ δεν είπαμε ότι το μόνο σημαντικό ζήτημα είναι να παραδίδονται όσο το δυνατόν περισσότερα δέματα, ανεξάρτητα από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Ε, απλώς θέλουμε μία, ένα, υπηρεσίες πιο προσιτές, πιο ευέλικτες, πιο ποιοτικές, ε, που μπορούν να, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της συνεργασίας. Πολλά μέρη της διαδικασίας μπορούν να βελτιωθούν χωρίς απαραίτητα να γίνει αυτό ε, σε βάρος των ε, εκείνων που βρίσκονται στο τέλος ε, της αλυσίδας παράδοσης των δεμάτων. για τη συνεργασία σας και αναμένω με χαρά μια πολύ επικοδομητική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νταντάν, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι κύριε Πρόεδρε, έλαβα την πρόταση. Ε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Θα το προτείνω λοιπόν απόψε το βράδυ για να μεταβάλουμε την συμβιβαστική μας πρόταση και νομίζω πρέπει να δεχτώ συγχαρητήρια από εσάς κύριε Πρόεδρε μέσα σε 12 λεπτά. Κύριε Νταντέν είστε ο ήρωάς μου, σας βεβαιώνω, πραγματικά. Να θυμίσω ε, ότι θέτεται ένα πολύ καλό παράδειγμα που θα έπρεπε να το ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Η ψηφοφορία είναι αύριο. Ε, τον Ιανουάριο είναι η ψηφοφορία στην Ολομέλεια και το Δεκέμβριο στην ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ. Στη συνέχεια τροποποίηση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών να πω ότι πριν δώσω το λόγο ότι η ψηφοφορία για τα δικαιώματα των επιβατών ε, είναι στις 17 Δεκεμβρίου. Ο λόγος είναι ότι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες δεν είναι εδώ σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, πράγμα που μας δίνει λίγο παραπάνω χρόνο. Ε, ο κύριος Μπάχα συμφώνησε γιατί προσπαθεί να επεξεργαστεί κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις από τις 566 τροπολογίες τις οποίες προσπαθεί να κεφαλώσει. Ε, και έχουμε τροπολογίες ε, ε, από συντάκτες που είναι τόσο διαφορετικοί, έχουν τόσο διαφορετική στάση. Μερικοί είναι ερωτευμένοι με τις αεροπορικές εταιρείες, άλλοι θέλουν να λιντσάρουν τις, ευρωπαϊκ, τις αεροπορικές εταιρείες. Κύριε Μπάχα, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε οι συνάδελφοι έχουν <laughs> ήδη ε, άγχος λόγω της καθυστέρησης ε, για την ε, έναρξη της συζήτηση και θέλουν αποζημιώσεις. Όπως είπατε το Δεκέμβριο θα γίνει η εξέταση για το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε περαιτέρω για το θέμα αυτό και να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε καλύτερες συμβαστικές λύσεις για τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Η δική μου θέληση είναι, ήταν να μπορέσουμε παρά τις δυσκολίες να φέρουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί στην τρέχουσα θητεία. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το Μάιο του 2014. Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες συνδέονται με το θέμα αυτό. Γιατί θα έχουμε και δυσκολίες αν δεν καταλήξουμε σε μια απόφαση. Όπως είπατε είναι πάνω από 500 τροπολογίες, αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των τροπολογιών ε, νομίζω ότι υποστηρίζει τη δική μου γραμμή. Όχι να λιντσάρουμε δηλαδή τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά να ξανατοποθετήσουμε σε πιο ισορροπημένο επίπεδο την πρόταση της Κομισιόν. Η βασική ιδέα θα ήταν να η κύρια ιδέα των τροπολογιών υποστηρίζει αυτό το οποίο εγώ έχω προτείνει. Θέλουμε να πείσουμε τις αεροπορικές εταιρείες να αλλάξουν γνώμη για ορισμένα θέματα και να καταλήξουμε σε κάποιες νέες καινοτομίε. Υπήρξε μια εταιρεία χαμηλού κόστους η οποία θα ήθελε όταν υπάρχει κάποιο σφάλμα στην κράτηση, παραδείγματο χάρη τυπογραφικό, να διορθώνεται αυτό. Αυτό δείχνει ότι αρχίζουν οι εταιρείε κάπου να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να έχουν μια άκαμπτη στάση εναντίον των επιβατών και να συνεχίσουν <clears throat> αυτό το οποίο κάνανε μέχρι τώρα. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν και σε προετοιμασία συμβαστικών τροπολογιών. Είχα επαφή με τους περισσότερους ε, σκιώδεις συγητές, θα ξαναβρεθούμε τη Δευτέρα και πιστεύω παρόλα αυτά την ευκαιρία να συζητήσουμε εδώ μερικά θέματα. Το θέμα της παροχής ε, αποζημιώσεων και υπηρεσιών μετά από μια καθυστέρηση βασί των άρθρων 6 και 7. Εδώ ήθελα εγώ να εξασφαλίσω μια κάποια ε, απλοποίηση στα χρονικά όρια που είχε θέσει η Κομισιόν, είχε πει 5, 9 και 12, εγώ λέω 3 και 5 ώρες μονάχα σαν όρια. Εδώ υπάρχουν βέβαια πολλές τροπολογίες των συναδέλφων σε σχέση με τα χρονικά αυτά όρια, πέρα από τα οποία θα πρέπει να υπάρχει κάποια παροχή υπηρεσία ή αποζημιώση. Και εδώ μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητούμε για τα θέματα αυτά. Ένα άλλο σημείο είναι το σημείο 4, όταν υπάρξει overbooking. Ο κύριος Ρικέ είχε καταθέσει μια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των άλλων. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου αναφέρεται η πολιτική του no-show ότι πρέπει να γίνεται όταν κάποιο δεν εμφανιστεί για επιβίβαση στην πτήση. Η δική μου θέση ήταν ότι πρόκειται για μια σύμβαση παροχής υπηρεσίας και επομένως δεν πρέπει να αρνείται η αεροπορική εταιρεία την πτήση επιστροφής για κάποιον ο οποίος δεν έχει παρουσιαστεί στην πτήση ΑΛΕ. Αλλά και αυτό είναι ανοιχτό σε συζήτηση με τους συναδέλφους. Ένα άλλο σημαντικό σημείο σε ό,τι αφορά τις έκτακτες περιστάσεις το που αναφέρεται στο άρθρο 2. και εκεί θα, πρέπει να προσαρτηθεί ένας κατάλογος σε παράτημα για το ποιες είναι οι έκτακτες περιστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επίσης υπάρχει μια πρόταση η οποία μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτός ο κατάλογος να γίνει επί τη βάση εξου, κατεξουσιοδότηση πράξεων, να τον κάνει αυτό τον κατάλογο η Κομισιόν, αλλά Θέλω, όπω είπαν και οι συνάδελφοι από την, ΜΚΟ, από ΙΜΚΟ, αυτός ο κατάλογος να είναι όσο το δυνατόν πιο εξαρτητικό και μονάχα στη συνέχεια, εάν χρειαστεί, η Κομισιόν να το συμπληρώνει. Το κόστος ε, στέγασης σε ξενοδοχεία των επιβατών σε έκτακτες περιστάσεις, το άρθρο 9 παραγραφός 4 και εδώ υπήρξαν πολλές προτάσεις για περιορισμό μέχρι τρεις νύχτες 100 ευρώ ή 80 ευρώ όταν υπάρχει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που πρέπει να στεγαστεί ο επιβάτης. Και εγώ θέλω να υπενθυμίσω την πρόταση της ΙΜΚΟ που προτείνει να υπάρχει ένα πλαίσιο 50 με 150 ευρώ. Βλέπετε ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα Και εδώ θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση. Σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας μιας εταιρείας, ήδη από το 2009 το Κοινοβούλιο είχε τονίσει την ανάγκη να υπάρξει μια αρρύθμιση και εδώ η πρόταση της Κομισιόν είναι υπερβολικά ήπια και αποδυναμωμένη και εδώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένας ε, δεσμευτικός κανόνας ο οποίος θα θεσπιστεί και περιμένω να ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων ε, σχετικά. Αυτά προς το παρόν τα κύρια σημεία τα οποία εγώ θα ήθελα να εγείρω και περιμένω με αδημονία τη συζήτηση με τους συναδέλφους που είναι παρόντες. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Σάβησα έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία, το πνεύμα συνεργασίας που έχει δείξει με τους σκιώδεις εισηγητές. Τα θέματα των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών εταιριών είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα, οδηγεί σε μια συναισθηματική αντιμετώπιση πολλές φορές και αυτό μπορεί να εξηγήσει και το μεγάλο αριθμό των τροπολογιών. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στον ε, ε εισηγητή και στους σκιώδεις εισηγητές. Έχουν πάρα πολύ έργο το οποίο θα πρέπει να κάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις 566 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Ο σκιώδης μας συγητής ε, για την ομάδα του, των φιλελευθέρων και εγώ ίδια πιστεύουμε ότι θα μπορέσει αυτό να δικήσει σε ένα εξισορροπημένο έγγραφο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των επιβατών την κατάσταση των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών. Όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο κείμενο ώστε να είναι χωρίς αμφισημίες και κατανοητό από όλους. Πιστεύω ότι οι επιβάτες θα πρέπει να γνωρίσουν και καλύτερα ποια είναι τα δικαιώματά τους από τη στιγμή που αγοράσουν ένα εισιτήριο μέχρι να τελειώσει το καθήκοντό το ταξίδι τους. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν ποιε είναι οι υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά τους. Αυτό δίνει μεγάλη εξουσία σε αεροπορικές εταιρείε. Φυσικά δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανισότητες μεταξύ των δικών μας αεροπορικών εταιρεών και των αεροπορικών εταιρεών σε άλλα μέρη του κόσμου. Υπάρχουν παρόμοιες τροπολογίες από πολλούς για την καθυστέρηση και τις αποζημιώσεις και εδώ θα πρέπει να βρούμε μια συμβαστική λύση η οποία να λάβει υπόψη τα, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους επιβάτες αεροπορικών εταιριών. Δεν πρέπει επίσης να παραβλέψουμε και τα συμφέροντα των περιφερειακών μας αεροπορικών εταιριών. Εγώ παραμένω Διαθέσει μια συζήτηση για συμβαστικές τροπολογίες και τονίζω επίσης ότι χρειαζόμαστε να εξασφαλίσουμε καλύτερα δικαιώματα για τους επιβάτες Λόγω περιορισμένου χρόνου βέβαια εγώ δεν πρόκειται να διεξέλθω όλες τις τροπολογίες μας σε λεπτομέρεια. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια θετική συνεργασία με τον εισηγητή και θα βρούμε μια λύση. Κύριο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Μπαχ, για την καταπληκτική δουλειά, ε, την οποία ελπίζω να εξελίξετε και περισσότερο. Αναφέρατε ε, στα αρχικά σας σχόλια την ανάγκη για την εξέβρεση μιας ισορροπίας. Δεν θα μιλήσω για όλες μου τις τροπολογίες, αυτό θα σας χαροποιήσει βέβαια, αλλά κυρίως για μια τροπολογία, την 8 η οποία προσπαθεί να επαναφέρει αυτή την ισορροπία. Ε, θέλει να υπάρχει να υπέχει ευθύνη η αεροπορική εταιρεία ε, από την σύμβαση που έχει συνάψει με τον καταναλωτή, με τον επιβάτη. Σε λίγε, όπως και σε ελάχιστες άλλες συναλλαγές, ο πελάτης πληρώνει εκ των προτέρων για την υπηρεσία. Πληρώνει καλόπιστα και προσδοκά ότι θα λάβει την υπηρεσία. Να πούμε τώρα ότι η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αποφύγει την, την ε, ικανοποίηση του συμβολέου, της σύμβασης, νομίζω ότι είναι κακή κίνηση. Άλλα στοιχεία της τροπολογίας, των τροπολογιών μου. Φυσικά υπάρχει το θέμα των ε, έκτακτων συνθήκων ή εξαιρετικών συνθήκων. Ε, με την τροπολογία μου προτείνω να υιοθετήσουμε τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, οι περιστάσεις θεωρούνται έκτακτες, εξαιρετικές, όταν δεν, μπορούν να αποφευχθούν, όταν δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, ακόμα και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Δηλαδή πρόκειται για περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου της αεροπορικής εταιρείας. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριό μας έβγαλε έναν πάρα πολύ καλό ορισμό και δεν πρέπει εμείς τώρα να καθίσουμε να ορίσουμε τι αποτελεί ή δεν αποτελεί έκτακτη εξαιρετική περίσταση. Ε, νομίζω ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί επί των κριτηρίων. Το θέμα της αποζημίωσης. είχαμε κάποιες πολύ ανησυχητικέ ε, ε, συναντήσεις με κάποιους Αυστριακούς οι οποίοι έχουν μία υπηρεσία παρακολούθησης των αξιώσεων των σχετικών με τις αεροπορικές εταιρείες και οι οποίοι μας είπαν ότι αν υιοθετηθούν οι προτάσεις της Κομισιόν, ένας μεγάλος αριθμός των αξιώσεων αυτών ε, δεν θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν. Είμαστε μεταξύ 3 και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, ε, ποσό το οποίο δεν θα καταβάλουν οι αεροπορικές εταιρείες στους επιβάτες. Ε, δεν θέλουμε οι αεροπορικές εταιρείες να υποφέρουν ανέτεια, αλλά, δεν, αλλά θέλουμε να υπάρχει και σωστή αποζημίωση των επιβατών. Το άρθρο 1, οι τροπολογίες του άρθρου 1 ε, θέλουμε ένα νέο προφίλ των ε, αξιώσεων αποζημίωσης, μια ε, επανεπεξεργασία του περιεχομένου των αξιώσεων αποζημίωσης. Θα θέλαμε καθυστερήσεις της μίας ώρας να φέρουν αποζημίωση ενός συγκεκριμένου αριθμού ευρώ και κάθε επιπλέον ώρα να επιφέρει μια επαύξηση. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 5 ώρες, θα πρέπει να προστίθενται 200 ευρώ. Ε, μάλλον αν είναι 5 ώρες 200 ευρώ και αν υπερβαίνουν τις 5 ώρες καθυστέρησης 500 ευρώ. Είναι περισσότερο τροφή για σκέψη ίσως, αλλά είναι και ένας δίκαιος τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει η πρόταση της Κομισιόν, πολλοί άνθρωποι θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Και δεν νομίζω ότι είναι η δουλειά του Κοινοβουλίου να θέτει τους πολίτες σε μειονεκτική θέση, τους ταξιδιώτες σε μειονεκτική θέση. Και τέλος, για την αιωτιολογικη σκεψη σκέψη 18α, όπου ζητούμε από τις αεροπορικές εταιρείες να παρέχουν ε, ε, συσκευές οξυγόνου δωρεάν για όσους τις χρειάζονται. Ζητούμε για ανεξάρτητη διαμεσολάβηση ε, για την επίλυση διαφορών μεταξύ ταξιδιωτών και αεροπορικών εταιριών. Και τέλος, υπάρχει η τελογική σκέψη 29 για, τον, για εξοπλισμό που θα πρέπει να μεταφέρεται στην καμπίνα. Δεν ξέρω, με, δεν ξέρω πόσα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνετε εσείς. Ε, εγώ όμως λαμβάνω ένα σωρό μηνύματα για το μουσικό εξοπλισμό. Ε, περιμένω με χαρά τη συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές και αναμένω τη σχετική συζήτηση με πνεύμα αισιοδοξία. Η κυρία Φώστερ. Thank Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας ε, τον κύριο Μπαχ. Ξέρω ότι διαφωνώ με κάποια τα οποία λέω εγώ, αλλά έχει κάνει τρομερή δουλειά. Γιατί είναι πολύ πολύ το θέμα αυτό. Από τις τροπολογίες μου το πιο σημαντικό είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πάει πουθενά εάν δεν ε, υπάρξει και μνήα τροπολογία που λέει ότι πρέπει να εφαρμόζονται όλα αυτά και στο Γιβραλτάρ γιατί και αυτό είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής όπω όπως αναφέρθηκε στη Συμφωνία του 2006. Αυτό τώρα για τα νομικιστικά. Επανέρχομαι τώρα στο, στην ουσία του θέματο. Νομίζω ότι έχω καταθέσει κάποιε επικοδομητικέ τροπολογίε. Συμφωνώ με πολλά από τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν από το έγγραφο, μέσα στο έγγραφο τη Κομισιόν, όπω ξέρει και η Κομισιόν, υποστηρίζουμε να κινηθούμε στα, στις 5 ώρες ως όριο για την αποσημείωση. Πιστεύω ότι η Κομισιόν της έχει δει τις τροπολογίες αυτές και έχουμε πει και κάποιες τροπολογίες πάλι επικοδομητικές για το ελάχιστο για την, για αποσημείωση σαν συνάρτηση του ελάχιστου κόστους των εισιτηρίων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι επικοδομητικά τι πρέπει να αποφασίσουμε τελικά. Εγώ έρχομαι από αυτό το χώρο και ξέρω ότι η παροχή υπηρεσιών είναι το κεφαλαιόδες. Αν δώσει, δεν δώσει κανείς τις απαραίτητες αυτές τις υπηρεσίες, θα πάει κάπου αλλού. Και νομίζω ότι οι αεροπορικές μας εταιρείες στην ε, Ευρώπη λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και καταφέρουμε να ερχόμαστε στο Κοινοβούλιο όταν χρειάζεται ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες το χειμώνα, θα μας φέρνουν εδώ οι εταιρείε. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Κύριε Τέιλορ, η κυρία Λίχτεμπερκ αναφέρθηκε σε κάποια στοιχεία, έτσι, δεν, είναι, δεν είναι παρούσα αυτή τη στιγμή εδώ. Ε, δεν ξέρω σε ποια χώρα αναφερόσασταν, αν ήταν η Αυστρία ή κάποια άλλη. Αλλά να ξαναγυρίσω υπάρχουν ακόμα θέματα που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση των ορίων 5, 9 και 12 ωρών. Αν έχουμε καθυστερήσεις οι οποίες μεταφέρονται από τη μία πτήση στην άλλη, μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα και αυτό το ξέρει και η Κομισιόν. Και πρέπει να δείτε και το αρνητικό αποτέλεσμα στην ε, χρήση πτήσεων από διαφορετικές εταιρείες αν πρέπει να πάει κανείς σε ένα αεροδρόμιο και να έχει μια ανταπόκριση, αυτό θα έχει νόημα. Δεν θέλουμε λοιπόν να εμποδίσουμε τον κόσμο από το να χρησιμοποιεί διαφορετικές εταιρείε. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λογικά. Σε σχέση με το να έχει η Κομισιόν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει της ε, κατεξουσιοδότησης πράξη για τις έκτακτες περιστάσεις, μα και εγώ μπορώ να σας πω ποιες είναι κατά τη δική μου άποψη οι έκτακτες περιστάσεις. Δεν πρέπει αυτό να είναι κάτι που αποφασίζει μόνο η Κομισιόν. Είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό, δεν είναι τόσο απλά. Υπάρχει φυσικά η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων που μπορούν να αποτελούν μια έκτακτη κατάσταση ή όχι. Είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα αυτό. Νομίζω ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προσπαθήσει να καταλήξουν σε ένα έγκυρο κατάλογο με τον οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε. Πρέπει να δούμε και ποια είναι τα σημεία τα οποία αναγνωρίζονται διεθνώ σε σχέση με τι έκτακτε περιστάσει και ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε συμβαστικέ λύσει. Νομίζω ότι είναι πολύ πλοκό το θέμα αυτό. εκατοντάδε τροπολογιών πρέπει να αντιμετωπίσει ο εισηγητή. Θα δούμε λοιπόν πώ θα πάνε τα πράγματα και θα δούμε ποια είναι η τελική θέση του εισηγητή και μπορούμε να καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίε αλλά είναι πολύ εύκολο να ρίχνουμε το φταίξιμο σε κάποιον άλλο, σε αεροπορικές εταιρείε. Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι μας έχουμε να εκπροσωπήσουμε <clears throat> τους ε, εκλογείς μας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αλυσίδα τροφοδοσίας των αεροπορικών εταιριών και επίσης και αυτούς που ωφελούνται όπως είναι ο τουρισμός. Θέλω λοιπόν να κλείσω εδώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πρόεδρε. Η κυρία Βερνιό, η σχεδόν συγκεκριά μας, δεν μπορεί να είναι εδώ, οπότε θα την ε, αντικαταστήσω. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπακ, τον εισηγητή, για την εξαιρετική του έκθεση. Πολλές τροπολογίες έχουν υποβληθεί. Αυτό βεβαίως δείχνει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί το σημαντικότατο αυτό ζήτημα. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τι τροπολογίε που πετυχάνουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των επιβατών και την αποτελεσματικότητα τη υλοποίηση των μέτρων θα πρέπει να ε, ξεκρυπωθούν περιττέρω και άλλοι ορισμοί νομοθετικοί για να, έχουμε, να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει νομική ασφάλεια και να καλύπτονται και οι επίγουσε καταστάσει, καθώ και η τιμή του εισιτηρίου θα πρέπει να καλύπτει εξ αρχή τι αποσκευέ που αποστέλλονται για φόρτωση ώστε να προστατεύονται όσο το δυνατόν καλύτερα οι επιβάτε. Επίση, η ε, ανάληψη πτήσης από υπεργολάβου υπεργολάβους από τρίτες εταιρείες θα πρέπει να καλύπτονται σε αυτές τις περιπτώσεις εφόσον δεν έχει ενημερωθεί ο επιβάτης και εφόσον υπάρχουν τρίτες χώρες που έχουν δικούς τους μεταφορείς ή η νομοθεσία είναι λιγότερο επωφελής για τον επιβάτη. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, αλλαγής μέχρι 48 ώρες πριν την πτήση με την, με την καταβολή ενός αντιτίμου και την περίπτωση του no-show, της μη ε, παρουσίας θα πρέπει να γίνει όπως ε, είπε η Μπερναντέτ μια εναλλακτική πρόταση. Θα πρέπει να υπάρχουν τρία στάδια, ε, διότι το τρίωρο για τα 450 χιλιόμετρα μου φαίνεται αδύνατο να γίνει σεβαστό. Τρία στάδια λοιπόν για τα 1500 μάλλον ε, χιλιόμετρα ε, και 7 ώρες για τα 1500 χιλιόμετρα και πάνω και για το 5000 χιλιόμετρα 10 ώρες. Βεβαίως μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά τα χρονικά όρια, αλλά επί της ουσίας θα πρέπει να βρούμε ε, μια μεσιωδό που να είναι υλοποιήσιμη. Ε, για την στέγαση τώρα. Οι τρεις πρώτες νύχτες που είναι πλέον σημαντικές θα πρέπει να καλύπτονται γιατί είναι και πιο συχνές περιπτώσεις χωρίς ε, όριο στην τιμή. Έπειτα θα πρέπει να υπάρχει ένα το όριο όπως 80 ευρώ ε, για την βραδιά αλλά για την πρώτη νύχτα ή τις δύο πρώτε τρεις πρώτε νύχτες θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτό νομίζω μπορούμε να το επεξεργαστούμε. Άρα, για τα όρια, τα χρονικά όρια των προσφυγών θα πρέπει να δούμε το τρίμηνο που αναφέρει ο κανονισμό ή το εξάμηνο σε κάποιε περιπτώσει για να υπάρχει επαρκή χρόνο και έπειτα, για να μην υπάρχει μεγάλη στρέβλωση του διαγωνισμό μεταξύ των κρατών Η σκιώδη ψυχητριά μα προτείνει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει έκθεση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν λάβει οι εθνικοί φορεί ω τώρα. Και εφόσον υπάρχουν μεγάλε αποκλήσει, να προτείνουμε μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Αυτά ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. De Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ιστορικό των δικαιωμάτων των επιβατών είναι μια μακρά ιστορία που ξεκίνησε με την έκθεση, τροπολογι... πρωτοβουλίας του κυρίου Τέιλορ που ανάγκασε την Κομισιόν να λάβει υπόψη όλα αυτά τα θέματα και στη συνέχεια η Κομισιόν είχε, έτεινε ευήκο ους και παρουσίασε μια έκθεση που γενικά αντιμετωπίζεται θετικά και νομίζω ότι και ο εισηγητής έχει καταφέρει να την βελτιώσει. Του μένει βέβαια ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο για να μπορέσει να συναρμόσει όλες αυτές τις τροπολογίες, αλλά το βασικό πνεύμα μας είναι σαφές. <clears throat> να δώσουμε έμφαση στα δικαιώματα των επιβατών και όχι στα δικαιώματα των εταιριών και των άλλων παικτών που βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Η Κομισιόν και αυτή προσπάθησε να εξασφαλίσει μια ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των θεμητών συμφερόντων. Αλλά εμεί τώρα θέλουμε να τονίσουμε πολύ περισσότερο τα δικαιώματα των επιβατών και όχι τις υποχρεώσει του. Όλοι οι τομείς όπου είναι δέσμοι οι καταναλωτέ παροχή τέτοιου είδου υπηρεσιών δεν θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα να αλυσμονούν οι εταιρείε τα συμφέροντα των επιβατών. Οι επιβάτε είναι καταναλωτέ αλλά είναι και πολίτε. Πρέπει να εξασφαλίζονται τα δικαιώματά του. Γι' αυτό είναι πολύ θετική η έκθεση του εισηγητή και αξίζει την υποστήριξή μα. Εγώ προσωπικά την υποστηρίζω ολόψυχα. Έχω καταθέσει δύο τροπολογίε που νομίζω ότι <clears throat> συνάδουν με το πνεύμα του εισηγητή και μπορούν επίσης να συμφωνήσουν και με άλλες προτάσεις ε, άλλων συναδελφών η 507 ότι θα πρέπει να αναφέρεται από τις εταιρείε ο όγκος και ο αριθμός των ε, ε, αποσκευών και επίσης η δυνατότητα να μπορούν να φέρουν στην καμπίνα του αεροπλάνου τα αγαθά που έχουν αγοράσει από καταστήματα duty free. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία νομίζω ότι τα δέχεται ο εισηγητής. Τώρα το θέμα του Γιβραλτάρ, κυρία Φώστερ, η οποία είναι ιδιαίτερα κομψή και στον τρόπο που μιλάει εξάλλου, δεν θέλησε να μπει καθόλου σε αυτή την πραγματική διαμάχη που υπάρχει μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου και ελπίζουμε όλοι ότι με το διάλογο θα μπορέσει να καταλήξει σε μια αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία και να τη σταματήσουν τα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά τούτου λεχθέντος αυτό το οποίο δεν είναι δυνατόν είναι να δεχτούμε αυτά τα οποία λέει η κυρία Φώστερ και ο κύριος Βάτσον να διαγραφεί η Συμφωνία του Λονδίνου του 1987. Και αναφέρεται εκεί ότι παραμένει εκκρεμής η κατάσταση του αεροδρομίου του Γεβραλτάρ μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία των δύο πλευρών. Η, <clears throat> Ισπανική κυβέρνηση με τη διακήρυξη της Κόρδοβας έχει καταγγείλει αυτή τη συμφωνία του 1987 και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ε, αντιμετώπιση που θα δώσει, τα, θα δώσει τη λύση στους νομομαθείς για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση στα θέματα αυτά. Αλλά μέχρι τότε εμείς παραμένουμε στο status quo όπως κάνει και η Κομισιόν και φυσικά ελπίζουμε ότι ο διάλογος θα μπορέσει σε φιλικό επίπεδο μεταξύ δύο χώρων που είναι και οι δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μια μακρά ιστορία θετικών και φιλικών σχέσεων να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή τη διαμάχη και να μην υπάρχουν και περαιτέρω <clears throat> επεισόδια μεταξύ των δύο χωρών. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς μας γοητεύει το θέμα αυτό, γιατί όλοι μας είμαστε πολύ καλοί πελάτες των αεροπορικών εταιριών, έχουμε τις δικές μας εμπειρίες και τους δικούς μας μαύρους καταλόγους για αυτά τα οποία γίνονται από τις εταιρείε. Έχουμε τις εμπειρίες μας πετώντας προς τις ε, Βρυξέλλες Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Ξέρουμε να, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη μεγαλύτερη κινητικότητα στις πτήσεις. Ο Μπαχ νομίζω έχει προσπαθήσει να ενισχύσει τα δικαιώματα των επιβατών εναντί της πρότασης της ε, Κομισιόν. Δεν συμφωνώ 100% αλλά θεωρώ ότι πάρα πολλά από αυτά που λέει είναι πολύ θετικά γιατί θέτουν στο επίκεντρο τον επιβάτη και όχι της επιχείρησης. Είχα δύο περιπτώσεις που εγώ προσπάθησα να εφαρμόσω τα δικαιώματά μου εναντίον των εταιριών. Μπορώ να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πολύ δύσκολη η, η θεραπεία των προβλημάτων που δημιουργούνται. Είναι πολλέ πολλές περιπτώσει. περιπτώσεις. Ένα είναι σαφές. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των εμπορικών αναγκών των εταιριών. Θέλουμε όλοι να έχουμε Ανταγωνιστικέ εταιρείε στην Ευρώπη, αλλά πρέπει και τα συμφέροντα των επιβατών να ληφθούν υπόψη. Κατά την άποψή μου λοιπόν η πρόταση τη Κομισιόν δεν είχε τη σωστή ισορροπία και νομίζω ότι η πρόταση του Τζορτ Μπαχ έχει βελτιώσει αυτή την ισορροπία γιατί εξασφαλίζει καλύτερα τα δικαιώματα των επιβατών. Ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα είναι η πληροφόρηση το να υπάρχει σε κάθε αεροδρόμιο ένας συνομιλητής για τον επιβάτη γιατί πολλές φορές αυτό δεν λειτουργεί. Τέλος, να σας πω ότι για μένα είναι σαφές <clears throat> ότι η αποζημίωση όταν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ή ακυρώνεται μία πτήση δεν θα πρέπει να συνδέεται με το εισιτήριο. Δεν σημαίνει ότι αν πληρώνει κανείς ένα φτηνό εισιτήριο θα είναι φτηνή και η αποζημίωση. Και περιμένω να δω τι θα γίνει στην περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Κράμερ. Χωρίς μικρόφωνο. η δική μου ε, εντύπωση με τις αεροπορικές εταιρείες είναι ότι πολλές φορές έχουν στα χαρτιά σχέδια τα οποία δεν λειτουργούν. Ξέρουν ότι θα υπάρξει καθυστέρηση και αυτό οδηγεί στο να καθυστερεί ο επιβάτης. Μπράιαν, και εσύ περίμενε δύο ώρες στη Φραγκφούρτη, εγώ είχα κάτσει παραπάνω, τρει ώρες και τέτοια. Σε ζηλεύω λοιπόν γι' αυτό. Τελικά κάνουν τα κέρδη του στην πλάτη του επιβάτη οι επιχείρησει. Εγώ έπρεπε να πάω στο Βερολίνο κάποια στιγμή και ακυρώθηκε η πτήση μου. Δεν πήρα την απογευματινή και πήρα μια βραδινή πτήση μου, πήγε καθυστερημένα, αλλά πήρα αποζημίωση μόνο για την πρώτη ακύρωση. Αν το ήξερα αυτό θα είχα αλλάξει ήδη την ε, κράτησή μου. Και εγώ πέταξα από τη Βασιλεία πρόσφατα στο Βέλγιο με 970 ε, ευρώ εισιτήριο και έπρεπε να πληρώσω 60 ευρώ για τις αποσκευές μου. Και αυτό δεν το έλεγε πουθενά όταν έκλεινα ε, την, το εισιτήριό μου. Δεν μου έλεγε ότι μπορώ να πάρω μία βαλίτσα ή δεν μπορούσα να πάρω παραπάνω κτλ. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν καμιά σχέση με, την, με το τίμημα του εισιτηρίου. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουν αυτές οι καταχρήσεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνω καθόλου είναι ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι πρέπει να είναι τρεις ώρες το όριο της καθυστέρησης. Γιατί για το τρένο πρέπει να είναι μία ώρα και εσείς θέλετε πέντε ώρες για τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν ακολουθείτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ακολουθείτε την άποψη των ε, αεροπορικών εταιριών. Από εκεί ξεκινάτε. Επίσης το να υπάρχει ένας ουδέτερος διαιτητής. Να μπορεί κανείς να προσφεύγει Ούτε καν έχετε αναφέρει στην πρότασή σας την ιδέα να υπάρχει μια μορφή διαμεσολάβησης, να υπάρξει μια πίεση προς τις αεροπορικές εταιρείες. Γιατί δεν έχετε δεχτεί την ιδέα αυτή και μας αφήνετε εμάς να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. 5, 9 και 12 ώρες. Ωραία. Αλλά όταν πηγαίνω <clears throat> με το τρένο για κάθε καθυστέρηση δύο ωρών παίρνω μια αποζημίωση. Γιατί να υπάρχει μια τέτοια διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί διαφορετική αποζημίωση στα τρένα από ότι σε αεροπορικές μεταφορές. Μπορεί να φτάσω πέντε ώρες καθυστερημένος και δεν παίρνω τίποτα λοιπόν. Δεν υπάρχει η συμμεταχείριση. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης το να μπορεί κανείς να κάνει την πτήση επιστροφής όταν έχει χάσει την πτήση που πηγαίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι για μένα αυτονόητο και για τις ε, έκτακτες περιπτώσεις. Νομίζω ότι και αυτό είναι σαφές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν, όταν δεν υπάρχουν έκτακτες ε, περιστάσεις, δεν πρέπει, πρέπει να πληρώνει οι αεροπορικές εταιρείες. Ακολουθήστε λοιπόν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το να κάνει ένα σφάλμα ο πιλότος, να υπάρξει ένα πρόβλημα, αυτό δεν είναι έκτακτη κατάσταση. Το να βαράει κανείς τις αεροπορικές εταιρείες, όπως είπε η κυρία Φώστερ, όχι εμείς τις πληρώνουμε τις εταιρείες, δεν τις βαράμε. Θέλουμε απλώς να έχουμε τα ίδια δικαιώματα όπως έχουμε στα τρένα, να τα έχουμε και στα αεροπλάνα. Εντάξει. Ναι, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Στην Φιλανδία <laughs> είχα πει σε κάποιον έχετε προβλήματα. Όχι, λέει, έχουμε πέντε μήνες χιόνι το χρόνο στο αεροδρόμιο, αλλά λειτουργούν όλα. Μια χαρά. Λοιπόν, πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να πούνε κάτι αντίστοιχο. <laughs> Άλλες χώρες δεν έχει, σε άλλες χώρες δεν έχει χιονίσει ποτέ τα τελευταία 30 χρόνια και παρόλα αυτά έχουν καθυστερήσει, τελευταίο σημείο που θέλω να πω τα μουσικά όργανα. Όταν θέλει κανείς να μεταφέρει μουσικά όργανα. Βέβαια δεν κυκλοφορεί κανείς με ένα μικρό φλάουτο τσέπης. Κυκλοφορούν με κοντραμπάσα και γκρανκάσες πολλές φορές. Υπάρχουν φοιτητέ μουσικής οι οποίοι πρέπει να ταξιδέψουν. Λοιπόν, και επίσης για το ποδήλατο. Άμα θέλει κανεί να πάρει ένα ποδήλατο, αυτό 90% των περιπτώσεων γίνεται. Λίγε εταιρείε αρνούνται να πάρει κανεί ένα ποδήλατο και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ καλό. Αν λύσετε το πρόβλημα τη μεταφορά ποδηλάτο, κύριε Μπαχ, θα σα αγαπώ πάρα πολύ και θα είμαι πάρα πολύ σύμφωνο μαζί σα. <coughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς όταν άκουγα τον κύριο Κράμερ να μας λέει πόσο του κόστισε το αεροπορικό του εισιτήριο και η βαλίτσα του. Δεν μας είπε πόσο του κόστισε να, να πάρει το ποδήλατό του στο αεροπλάνο. Ε, ε, ε, αναρωτιόμουν να θα μας δώσετε λεπτομέρειες για το κόστος. Τέλο πάντων, υπάρχουν πολλέ τροπολογίε οι οποίε έχουν να κάνουν με την άμεση μετάφραση του κόστου από την έκθεση πρωτοβουλία του κυρίου Τέιλορ που την είχαν στηρίξει οι συνάδελφοι την τελευταία φορά. Και έχει να κάνει περισσότερο με του ε, αναπήρου και του ε, ανθρώπου με ιατρικέ ανάγκε και ε, με αναπηρίε. Εδώ ελπίζω να υπάρξει συνένεση για να προωθηθούν αυτά τα ζητήματα. Επίση, πρόεδρε, στι προκατακτικέ ερωτήσει που είχαμε για το όλο θέμα, έκανα και εγώ κάποιε παρατηρήσει για την ανάγκη να ενισχυθούν οι φορεί ε, οι εθνικοί φορεί επιβολή. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να επιβληθούν τα μέτρα ή να εξεταστούν οι αξιώσει των επιβατών, εφόσον υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετά ενδυναμωμένοι οι φορεί σε εθνικό επίπεδο για να μπορέσουν να ε, καλύψουν τι προσφυγέ που υποβάλλονται. Οπότε ελπίζω οι τροπολογίε μου να γίνουν δεκτέ για να οδεύσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Επίση, να συμπληρώσω την έκθεση του κυρίου Μπακ με τι τροπολογίε μου το επιδίωξα για να έχουμε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για τι έκτακτε συνθήκε. Συμφωνώ εδώ με την κυρία Φώστερ. Δεν πρέπει να δώσουμε κατάλογο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εμπιστευτούμε μέσω κατεξοσοδότηση πράξη. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο κατάλληλο τρόπο να προχωρήσουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε όμω οπωσδήποτε και μάλιστα σε νομοθετικό επίπεδο είναι νομική ε, σαφήνεια για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να είναι σαφέστατο για τον επιβάτη εάν έχει δικαίωμα για αποζημίωση ή όχι. Και αυτό φυσικά τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει. Και άλλε δύο σύντομε παρατηρήσει, Πρόεδρε. Πρώτον, ω προ την αποζημίωση όταν έχει παραμείνει σταθμευμένο πολλή ώρα σε ένα νεροδιάδρομο κάποιο αεροσκάφο. Για λόγους ασφάλειας πρέπει να δούμε εάν υπήρξαν υπόνοιες ε, ε, απειλής ή απειλές για την ασφάλεια. Η διάρκεια του τρίωρου νομίζω ότι είναι αρκετή για τον διάδρομο και για τις καθυστερήσεις εν γέννη. Δεν νομίζω ότι ότι θα ήταν παράλογο να καταβάλλεται από ζημίωση, μάλιστα για μικρή διάρκεια πτήση, για μια καθυστέρηση πάνω από τρίωρο. Νομίζω ότι είχε τοποθετηθεί σχετικά το Κοινοβούλιο και στη δική μου την τροπολογία προσπαθώ να αποκαταστήσω την αρχική μα ε, συνένεση. Διότι είναι πολύ δυσάρεστο σε σύντομε πτήσει εντό Ευρωπαϊκή Ένωση που κάποιε φορέ είναι και λιγότερα από μία μισή-δύο ώρε να υπάρχει τρίωρη καθυστέρηση. Δεν είναι παράλογο λοιπόν να πούμε ότι είναι αυτό το όριο για να αρχίσει να καταβάλλεται μετά αποζημίωση. Πάντω αυτό είναι λίγο πολύ, το, αυτή είναι η αιτιολόγηση των ε, τροπολογιών που υπέβαλε. Ο κύριο Μπένιον, ευχαριστώ πρόεδρε. Η παρατήρηση του κυρίου Κράμερ για τι αποσκευέ του. Εγώ ταξίδευα το όλη μου τη ζωή και πολύ θα ήθελα να επιδοτηθώ από τι αποσκευέ του κυρίου Κράμερ και όσα πληρώνει. Αλλά για να περάσω στην έκθεση αυτή καθεαυτή, ο κύριος Τέιλερ νομίζω είπε ότι είναι ζωτική σημασία να έχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των επιβατών και τις ανάγκες των ε, φορέων, των παρεχόντων των υπηρεσιών. Σωστό είναι αυτό, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Μην ε, υπερυθμίσουμε τον, ε, το όλο σύστημα, ώστε τελικά να είναι πιο επωφελές για έναν ε, παρέχοντα να ακυρώσει τελείως μια πτήση παρά να καθυστερήσει κάποιες ώρες. Ε, εφόσον κάποιες φορές υπάρχουν δύο πτήσεις καθημερινώς, θα πρέπει να φροντίσουμε να δίνουμε και επαρκή κίνητρα μέσω της νομοθεσίας μας. Τώρα για τις στάσεις ε, μεσοπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες. Θα συμφωνήσω με την τροπολογία του κ. Μπάτμπορν για το τρίωρο. Ε, αλλά είναι πολλές οι πτήσεις στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή με ταξιδιώτες που μπορεί να πάνε και να έρθουν μέσα στην ίδια μέρα. Εάν υπάρχει τρίωρη καθυστέρηση, ο λόγος ύπαρξης του ταξιδιού καταρρύπτεται. Δεν μπορεί λοιπόν να μην παίρνει κανεί καμία αποζημίωση μέχρι, να, ε, μέχρι την καθυστέρηση του, του, του πεντάωρα. Αν έχει χάσει τη συνάντηση για την οποία ξεκίνησε, είναι γελίο. Τρει ώρε νομίζω λοιπόν είναι εύστοχο για τι σύντομε διάρκεια πτήσει. Και πάλι όμω για αυτέ τι πτήσει η κατάσταση μπορεί να είναι τελείω διαφορετική. Σε άλλα μέρη του κόσμου ε, λίγε ώρε καθυστέρηση δεν σταματούν τον επιβάτη από το να ε, πραγματοποιήσει το ταξίδι του. Κάποιε φορέ ένα αεροσκάφο πρέπει να αντικατασταθεί και μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση αρκετών ωρών. Μερικέ φορέ και μισή μέρα. Είναι όμω διαφορετικέ συνθήκε. Εδώ μιλάμε για ιδιαίτερε ε, συνθήκες. Τώρα για τις ε, πτήσεις transit, τις ε, διασυνδέσεις δηλαδή, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί πραγματικά ε, λυπούμε για τους επιβάτες των οποίων η ανταπόκριση έχει καθυστερήσει. Την χάσανε γιατί η πρώτη άργησε. Παρόλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια σύντομη πτήση και μετά μια πιο μεγάλης διάρκειας. Ιδίως από τα μικρά τοπικά αεροδρόμια ξεκινώντας. Εάν συγκεντρώσουμε όλη την ευθύνη στον ε, υπεύθυνο για την σύντομη πτήση, θα καταλήξουμε να καταργήσουμε τα κίνητρα. Τα κίνητρα των εταιριών χαμηλού κόστου που αυτή τη στιγμή λειτουργούν και δεν θα καλύπτονται κάποιε ανταποκρίσει. Δηλαδή, κάποιε φορέ όταν παίρνει κανεί κάποιε σύντομε πτήσει, είναι σαν να αναλαμβάνει ίδιο τον κίνδυνο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε μία πτήση 1500 ευρώ ως προς την αξία, καμία ευθύνη και όλη την ευθυνά την αναλαμβάνουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την πτήση των 50 ευρώ. Νομίζω ότι ακόμα και η ε, Ryanair δυσκολεύεται με τον backroll, ε, αλλά οποιοδήποτε περιορισμός για τα προϊόντα, ε, τα δοσμολόγητα, τα duty free, θα πρέπει να είναι γνωστό αυτό τον επιβάτη. Τη στιγμή που κάνει την κράτηση και τη στιγμή που κάνει το τσακίν. Ακόμη και όταν αλλάζει πτήσει και ανακαλύπτει ότι πρέπει να περάσει πάλι από την ασφάλεια κάποιο και τα μπουκάλια που αγόρασε στο duty free μετά χρεώνονται στη δεύτερη πτήση. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να είναι γνωστά και ουσιαστικά εξαγριώνουν τον κόσμο και κάτι που αναφέρε ο κύριος Μπράτμπορν για τους ε, ανθρώπους με αναπηρίε. Όταν μια αεροπορική εταιρεία απαιτεί ο ε, ανάπηρος να συνοδεύεται από κάποιον φροντιστή, θα πρέπει και αυτός να γνωρίζει τι δασμοί ισχύουν στο αεροδρόμιο και πώ θα ε, κοστολογηθεί η παρουσία του. Και αυτά θα πρέπει να είναι γνωστά. Πρέπει να προβλεφθεί σχετικά και μια τροπολογία, νομίζω. Να σα θυμίσω ότι τα δασμολόγητα βέβαια και η καταβολή του δασμού ή όχι έχουν να κάνουν με τα εισοδήματα των εθνικών κυβερνήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ είμαι ο συντάκτη γνωμοδότηση από την Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και Καταναλωτών, ΙΜΚΟ. Γι' αυτό εμεί έχουμε δει και την οπτική γωνία του καταναλωτή στην Επιτροπή μα <clears throat> Έχω 237 ε, ε, τροπολογίες και 10 συμβιβαστικές. Θα ψηφίσουμε αύριο. Ελπίσουμε η δική μας πτυχή για την προστασία του καταναλωτή θα τύχει και ευήκοης ακρόαση από τη δική σας Επιτροπή. Κάποια λίγα σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μας. Πρώτα απ' όλα, η επιχειρηματολογία των των αεροπορικών εταιριών που λέει ότι άμα δεν πετάτε ακυρώνεται όλη η κράτησή σας, αυτό είναι κάτι που δεν το δεχόμαστε. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει αθέτηση συμβολέου. Επιχειρήματα όπως το no show ότι δεν εμφανίζεται κανείς, αυτά δεν μπορούμε να τα δεχτούμε και εδώ νομίζω μπορούμε να είμαστε σύμφωνοι. Η πρώτη συμβαστική τροπολογία αντιμετωπίζει τις έκτακτες περιστάσεις. Τι είναι αυτές οι περιστάσεις. Υπάρχει εδώ το παράρτημα το οποίο όμως πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια. Γι' αυτό η πρότασή μας είναι <clears throat> ότι αυτές είναι είναι περιπτώσεις <clears throat> οι οποίες είναι κατανοητές και σύγνωστες και αυτές οι οποίες δεν μπορούν να είναι σύγνωστες για τις αεροπορικές εταιρείες. Δηλαδή, άμα είναι ανέθυνη μια αεροπορική εταιρεία, δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί ότι είναι αποδεκτό. Αν, γίνει, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα λόγω ε, ελλειπούς ε, συντήρησης ενός αεροπλάνου ή ελλειπούς ε, συντήρησης εδάφους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο επιβάτης φταίει. Ο επιβάτης μπορεί να έχει μια αίτηση αποζημίωσης από τις εταιρείε εξυπηρέτησης, αλλά ο επιβάτης όχι. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να το μετακυλεί στον επιβάτη η αεροπορική εταιρεία. Αυτό λοιπόν η βασική μας <clears throat> αντιμετώπιση γι' αυτό προτείνουμε ένα κατάλογο ο οποίος είναι συγκεκριμένος, ο οποίος δεν είναι εξαρτητικός. Μπορεί η Κομισιό λοιπόν, εάν υπάρχουν περαιτέρω ε, έκτακτες περιστάσεις που κανείς από εμά δεν το έχει σκεφτεί, να συμπληρώσει εκεί στον κατάλογο. Μπορεί να προσθέσει, όχι όμως να αφαιρέσει ή να ακυρώσει έκτακτες περιστάσεις που περιλαμβάνονται στο παράτημα. Έτσι λοιπόν δεν ακυρώνεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πολιτική για τον νοσο, για την μη εμφάνιση, είμαστε σαφείς εδώ όταν ένας επιβάτης είτε είναι το αλέ, είτε είναι η επιστροφή, είτε είναι ένα κομμάτι μιας πτήσης πολλών, μιας, ε, ενός ταξιδιού με πολλές πτήσεις, ο καταναλωτής έχει πληρώσει για όλη την διαδικασία και όχι για ένα κομμάτι μονάχα. Η εταιρεία λοιπόν το έχει λάβει αυτό υπόψη. Αν δεν είναι παρόν και έχει πληρώσει γιατί θα πρέπει να πληρώσει ένα περαιτέρω τίμημα όταν δεν έχει πάρει το αεροπλάνο. Δεν πρέπει να υπάρχει κάτι περισσότερο. Απλώ η αεροπορική εταιρεία πρέπει να έχει το δικαίωμα μισή ώρα πριν, έρθει, πριν φύγει το αεροπλάνο, αν δεν είναι παρόν, να δώσει τη θέση του σε κάποιον άλλο. Καθυστέρησε τώρα στο Τάρμακ, στην πίστα του αεροδρομίου. Έχουμε ένα ε, μια συμφωνία που έχουμε, στην οποία έχουμε καταλήξει για το χρόνο στον οποίο θα πρέπει να αποβιβαστούν οι επιβάτες από το αεροδρόμιο, από το αεροπλάνο. Αλλά εάν τώρα πρόκειται το αεροπλάνο να φύγει στο τέλος αυτού του διαστήματος, αυτό βέβαια δεν έχει πολύ ε, νόημα, γι' αυτό αφήνουμε ένα περιθώριο μισής ώρας, ώστε να αποφασίσει ο πιλότος. Αν πει ο πιλότος ότι σε 10 λεπτά θα ξαναφύγουμε και σε 20 λεπτά, ε, μάλλον σε 10 λεπτά θα κινηθούμε από το διάδρομο και σε 20 λεπτά θα πετάξουμε, εκεί πέρα δεν έχει νόημα να αποβιβάσουμε τους επιβάτες επειδή έχει εκπνεύσει το όριο. Να υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο μισής ώρας για να υπάρξει προσαρμογή στην πραγματικότητα. Η πολιτική των ε, πληροφόρηση των επιβατών συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Το ίδιο πράγμα και για τις αποσκευές θα πρέπει να είναι σαφές στην αρχή της κράτησης να ξέρει ο επιβάτης τι κοστίζει αυτή η κράτηση και να περιλαμβάνει τα πάντα. Αλλά πρέπει να είναι απόλυτα σαφή αυτά τα στοιχεία και ποιο είναι το δεσμευτικό κόστος της πτήσης. Δεν μπορεί να λέει κανείς «Α, θα πληρώσετε με πιστοτική κάρτα, είναι άλλα 30 ευρώ». Αυτό πρέπει να αποκλείεται. τα αγαθά duty free. Πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνονται να πετάει κανείς με αυτά χωρίς πρόσθετη επιβάλληση. Θα αποφασίσουμε αύριο στο σημείο αυτό <clears throat> και για το Γιβραλτάρ. Εμείς θα βλέπουμε τα πράγματα από την πλευρά της ε, ασφάλειας των επιβατών. Και η Αγγλία και η Ισπανία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν παίζει, λοιπόν, δεν παίζει ρόλο ποιος έχει περισσότερο ή λιγότερο λόγο στον τομέα αυτό. Εφόσον οι επιβάτες κινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση. Δεν πρέπει να υπάρχει λοιπόν εξαίρεση. Αυτό είναι η δική μας θέση. Για το πώς θα ερμηνευτεί η Συμφωνία Αγγλίας και Ισπανίας. Και τώρα για το χρόνο αυτό που αναφέρεται για το κατόφλι της καθυστέρησης 3 ώρες, 5 ώρες. Νομίζουμε και εμείς δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω πολυπλοκή, περιπλοκή και θεωρούμε ότι έχουμε συνεργαστεί με τον κύριο Μπάχ, είναι πολύ καλή η δική του πρόταση, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων, δεν έχουμε μεγάλες διαφορές, νομίζω σε πάρα πολλού τομείς συμπίπτουν οι απόψεις μας. Ξέρετε, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τις ε, ε, ομαδικές πτήσεις και επομένως θα επανέλθουμε και στο ίδιο σημείο και ελπίζω να έχουμε πάλι επικάλυψη στα σημεία αυτά. Κυρία Σενέλοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάπως ε, βγήκα εκτός ε, του καταλόγου των αγορητών, αλλά ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο παρόλα αυτά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπακ για την εξαιρετική έκθεση που ετοίμασε. Και χωρίς να επαναλαμβάνει πράγματα που ήδη έχουν υποθεί εδώ από άλλους συναδέλφους, να επικεντρωθώ σε δύο μόνον τροπολογίες. Ε, που έχω υποβάλει εγώ η ίδια ή από κοινού με συναδέλφους. Η 219 κατά πρώτον για το άρθρο 2 σε ό,τι αφορά τους ορισμούς. Τους ορισμούς για την τιμή του εισιτηρίου. Ε, θα ήθελα να αποκλειστεί οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση προς την τιμή του εισιτηρίου από την αεροπορική εταιρεία βάσει της χώρας προέλευσης του επιβάτου. Η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου θα πρέπει να είναι ίδια, είτε αγοράζει κανείς το εισιτήριο από την Δημοκρατία της Τσεχίας, είτε από το Βέλγιο και η ίδια εφόσον το εισιτήριο είναι το ίδιο. Εξασφαλίζει την ίδια θέση, διότι δεν θέλουμε αδιαφανή ή διπλή ουσιαστικά τιμολόγηση της αεροπορικής θέσης. Είναι άδικο για τους αυτό δεν θα εξυπηρετήσει σε τίποτα ούτε την ε, ενίσχυση της κοινή αγοράς. Επίσης η 447 την οποία έχω αποβάλει από κοινό με τον κύριο Σίμψον. Είναι ένα νέο εδάφιο για το άρθρο 14, το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη να ενημερώνονται οι επιβάτες εφόσον υπάρχει απέτηση για το πού να απευθυνθούν οι επιβάτες, πού να ζητήσουν ε, βοήθεια. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να είναι σαφή, εύληπτα και ε, εύκολη πρόσβασή τους ταυτόχρονα με το εισιτήριο και με το boarding pass, διότι οι υποχρεώσεις του επιβάτη πολλές φορές αναφέρονται ευκρινώς, αλλά δεν είναι πολύ ενημερωμένοι οι επιβάτες συνήθως για τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα λοιπόν να με στηρίξετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ ίδιος, συνάδελφοι, να ξεκινήσω λέγοντας με το τι γίνεται με τα μουσικά όργανα. Μια φορά δεν μου επέτρεψα να πάρω το μπαστούνι μου του κρίκετ ε, στο αεροσκάφος μου είπαν ότι είναι ένα επικίνδυνο όπλο. Προφανώς οι περισσότεροι δεν με έχουν δει να παίζω κρίκετ. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται και με το μπαστούνι του κρίκετ πρέπει να φύγει πίσω στη σκευοφόρο γιατί θεωρήθηκε επικίνδυνο όπλο. Τέλος πάντων, για την ε, ανώτατη βία. Αυτό είναι η ουσία όλων των επιχειρημάτων. Σας θυμίζω ότι εδώ μιλάμε για νομοθέτημα που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, όχι της αεροπορικής εταιρείας. Κοιτάζοντας τις τροπολογίες, είδα πολλές, πολλές που με ανησύχησαν, διότι προσπαθώντας να συμβιβάσουμε την ανωτέρα βία με τα υπόλοιπα, τι θα δημιουργήσουμε, περισσότερα παραθυράκια για την ανώτερη βία από ό,τι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Για μένα λοιπόν οι έκτακτες αυτές περιστάσεις, η ανώτατη βία, θα πρέπει να είναι κάτι που να το διευκρινίσουμε πολύ προσεκτικά. Δεν θέλω ένα μακροσκελή κατάλογο, θέλω ένα συντομότατο κατάλογο για την ε, φως ε, μαζέρο όπως λέγεται, σε καμία περίπτωση τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στον ιστοτοπό τη έχει δημοσιεύσει κάτι που θεωρείται ως ε, το τελεσίδικο κείμενο από τις αεροπορικές εταιρείες, σε καμία περίπτωση δεν το θέλουμε αυτό. Και δεν θέλουμε καθόλου να πρέπει να βασιστούμε και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Διότι από την απόφαση τους ε, έχουν τελείως γλιτώσει οι αεροπορικές εταιρείες την αγνοούν, χρησιμοποιούν το επιχείρημα της της βίας και δεν πληρώνουν σε καμία περίπτωση αποζημιώσεις στους επιβάτες. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς και υπ' αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα κατάλογο κακό όπως είναι, ε, ως έχει και θα είναι χειρότερο με κατεξοδότηση πράξη. Αλλά να σα θυμίσω, συνάδελφοι, όχι τόσο καιρό πριν, πριν να μπαίνετε κάποιο Εσεί, εσεί εδώ, είχατε ξεσηκωθεί για την κατεξοδότηση πράξη, για τα δικαιώματα ε, σε σχέση με τα, με με το επιβατικό προσωπικό, με το προσωπικό τη πτήση, μάλλον. Και τώρα για τους επιβάτες θέλετε κατά εξοδότηση πράξη. Εγώ δεν τους εξοδοτούσα τίποτα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Διότι τα έχουν ε, κάνει σαλάτα και στο παρελθόν και ουσιαστικά τι θα του κάνουν, θα επιτρέψουν στις αεροπορικέ εταιρείε να πάρουν το κομμάτι τη νομοθεσίας που τους βολεύει και να κάνουν ό,τι του αρέσει. Όχι κατά εξοδότηση πράξη λοιπόν. Με ανησυχεί αυτό, αλλά όπω είπε και ο κ. Μπάνιον για του ε, αναπήρου και του ανθρώπου με μειωμένη κινητικότητα. Έχουμε ξεχάσει κάτι σημαντικό ε, στη βιασύνη μα αυτή για το τι θα πρέπει να αποκαλέσουμε αποζημίωση και πώς να καθοριστεί. Η ικανότητα, το δικαίωμα Τη κινητικότητα που χρειάζονται οι πολίτες, το δικαίωμα να πετάξει κανεί. δηλαδή. Έχει απόλυτα δίκιο ο συνάδελφος. Δεν τα πήγαμε καλά με αυτή την νομοθεσία. Ό,τι υλοποιηθεί την ερχόμενη φορά θα πρέπει να μπορούν να το ε, επιβάλλουν οι εθνικοί φορείς που για την ώρα έχουν αποτύχει τραγικά να το κάνουν για την κυρία Σενέλοβα. Τα δικαιώματα των επιβατών πρέπει να γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο που οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν δεν αναφέρουν πουθενά τα δικαιώματα του, του, επιβάτη. Αν είσαστε αρκετά μεγάλοι, θα θυμάστε αυτά τα ωραία, τα γυαλιστερά βιβλιαράκια που χρησιμοποιούσαμε, που Ανέφεραν το Μόνρεαλ, τη Βαρσοβία, όλε αυτέ τι συμβάσει και αυτή τη στιγμή τι έχει κανεί, έναν τεράστιο κατάλογο που δεν αναφέρει καμία πληροφορία για τα δικαιώματα του επιβάτη. Πιστεύω ε, σαφώς ότι η αποζημίωση θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει της ε, του προβλήματο που έχει δημιουργηθεί, όχι βάσει τη τιμή του εισιτηρίου. Διότι τι τιμή θα βάλει κανεί. δεν ξέρω, ε, στο αν έχασε κάποιο μια κηδεία στην οποία πρέπει οπωσδήποτε να πάει. Και μπορεί να έχει πληρώσει για το αρχικό εισιτήριο 50 ευρώ στην αεροπορική εταιρεία. Όχι, η αποζημίωση πρέπει να βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, αριθμό αναφοράς σε σχέση με την δυσκολία που δημιουργήθηκε στον επιβάτη. Και θα ολοκληρώσω με αυτό, συνάδελφοι. Όταν ήμουν δάσκαλο με ρώτησαν πώς μπορεί να βελτιωθεί κανεί στη δασκαλία. Και εγώ είπα, είναι τέλειο όταν δεν μπορεί, έχει κανείς να διδάξει σε παιδιά. Εάν ρωτήσει λοιπόν τι αεροπορικέ ε, εταιρείε πώ θα βελτιωθεί η αεροπλοεία, θα σα πούνε άμα δεν υπήρχαν επιβάτε. Μην ξεχνάμε λοιπόν ποιο είναι εδώ το, το κέντρο της προσοχής μας. Θα πρέπει να είναι επιβάτες και τα δικαιώματα των επιβατών. Και το επαναλαμβάνω, είναι μια οδηγία, ένα νομοθέτημα για τα δικαιώματα των επιβατών, όχι για τις αεροπορικές εταιρείες. Σας ζητώ λοιπόν συνάδελφοι, σας παρακαλώ θερμά, προσέξτε, είστε κάπως ήπιοι, κάπως ευγενικοί με τις αεροπορικές εταιρείες. Στις συμβιβαστικές σας ε, θα καταλήξουμε να έχουμε περισσότερες εκθέσεις τελικά από ό,τι ξεκινήσαμε να συντάξουμε. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί κατά την άποψή μου. Και Κύριε Καλαμίτσο. Thank you, thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την πίστη σας στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπαχ για την καλή και λογική του έκθεση και για τις πάνω από 500 τροπολογίες που υπέβαλαν οι βουλευτές. Πράγμα που δείχνει και το ενδιαφέρον του θέματος. Το κάτω-κάτω όλοι είμαστε επιβάτες. Αληθεύει ότι πολλές από τις τροπολογίες προσπαθούν να διευκρινίσουν τα δικαιώματα των επιβατών και να αυξήσουν την ασφάλεια δικαίου. Ωστόσο, ταυτόχρονα, αν, εξετάσετε, αν εξετάσετε προσεκτικά τις τροπολογίες, ε, φοβόμαστε ότι απομακρύνονται από τους στόχους που είναι η αναθεώρηση ε, των κανόνων για την επιβολή των δικαιωμάτων των ε, ε, επιβατών, αλλά και μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των επιβατών και του οικονομικού αντίκτυπου που έχουν αυτά τα μέτρα προστασίας ε, στις αεροπορικές εταιρείες και που έμεσα μετακυλίονται στους επιβάτες. Γιατί αν κλείνουν οι αεροπορικές εταιρείες και έχουμε μόνο αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους ή εταιρείες από τρίτες χώρες, οποίες τότε δεν μπορεί να διεκδικήσει κανείς επιβάτης ε, τα δικαιώματά του. Αυτά ήθελα να πω εν είδη εισαγωγή. Κάποια σχόλια τώρα που αφορούν τις περισσότερε τροπολογίε, Καθυστέρηση και αποζημίωση. Όπως εξηγήσαμε και σε προηγούμενες περιπτώσεις, το τρίωρο είναι ανεπαρκές. Ε, ανάλογα με τις αιτίες ε, της καθυστέρησης που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες ακυρώσεις. Το έχουμε δει αυτό. Εάν η αεροπορική εταιρεία πρέπει να, να πληρώσει ούτως ή άλλως μια αποζημίωση, είναι για αυτήν πιο συμφέρον να ακυρώσει την πτήση και να αυξήσει την καθυστέρηση, μεταφέροντας τους επιβάτες σε άλλες πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί ακόμα πιο αργά. Οι ακυρώσεις, θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι χειρότερες από την καθυστέρηση. Γιατί πάντοτε εξαρτάται η κατάσταση από το αν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις στις επόμενες πτήσεις, αν υπάρχουν επόμενες πτήσεις. Επομένως θα πρέπει πράγματι να συναρτάται η αποζημίωση με τις αιτίε της καθυστέρησης. Μετά έχουμε το ποσό της αποζημίωσης. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρήσει το ύψος της αποζημίωσης να το συνδέσει με την τιμή του εισιτηρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε ότι η αποζημίωση έχει να κάνει με την απώλεια χρόνου του επιβάτη. Δεν έχει να κάνει με την τιμή του εισιτηρίου. Τρίτον, Νομίζω πολύ το ανέφεραν. Οι εξαιρετικές, οι έκτακτες περιπτώσεις, οι συνθήκες. Αυτό που προτείνουμε νομίζω ευθυγραμμίζεται με την ομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Ε, δυστυχώς πολλές από τις προτινόμενες ε, τροπολογίες αποκλίνουν από, από την ομολογία των δικαστηρίων η Επιτροπή θεωρεί ότι ε, τεχνικά ελαττώματα που έρχονται στο φως ε, στη διάρκεια των ε, τακτικών ελέγχων δεν συνιστούν έκτακτες περιστάσεις. Ωστόσο, όταν έχει γίνει σωστά η επισκευή, η συντήρηση, τυχόν αναπόφευκτα και απρόβλεπτα τεχνικά ελαττώματα δεν θα πρέπει να οδηγούν σε αποζημίωση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ε, να αποφύγουμε την εμπορική πίεση επί των πιλωτών όταν πρέπει να λαμβάνονται ζωτικές αποφάσεις για την ασφάλεια της πτήσης και του αεροσκάφους. Τέταρτον, το περίφημο rerouting. Ε, ο εισηγητής προτείνει το δικαίωμα re-routing στους ε, επιβάτες των οποίων η πτήση έχει καθυστερήσει. Πρόκειται για ένα νέο δικαίωμα. Δεν υφίσταται με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο. Σε περίπτωση καθυστέρησης ε, θεωρείται ότι η πτήση θα, θα, θα γίνει. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση όπου ο επιβάτης μπορεί να πρέπει να μπει σε ένα άλλο δρομολόγιο ε, και να χρησιμοποιήσει την ίδια εταιρεία. Πράγμα που θα συνεπάγεται ίσως φοβερό κόστος και για τις δύο πλευρές. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν σε αυτή την περίπτωση του rerouting. Και τέλος κάτι που αναφέρθηκε νομίζω και στην προηγούμενη έκθεση, ο τρόπος αντιμετώπισης της διαμονής των επιβατών σε έκτακτες συνθήκες. Κατανοούμε ότι κάποιοι από τους βουλευτές θέλουν έναν πιο φιλικό προς τον καταναλωτή τρόπο διαμονής για τους επιβάτες. Εμείς προτείνουμε πράγματα που ισχύουν και με άλλους τρόπους μεταφορών, γιατί η απεριόριστη ευθύνη μια εσωροπορική εταιρείας για τους επιβάτες ε, για πράγματα που δεν ελέγχει είναι μια μοναδική περίπτωση, να μην το υποτιμούμε. Είναι κάτι που δεν υπάρχει σε άλλους οικονομικούς τομείς υπάρχει ο κίνδυνος επιβίωσης της αεροπορικής εταιρείας που έμεσα έχει αρνητικές συνέπειες για τους επιβάτες. Δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένες αναφορές για χώρες που είχαν τρεις αεροπορικές εταιρείες και τελικά κατέληξαν με μία μόνο αεροπορική εταιρεία και φυσικά ο, ο επιβάτης πληρώνει. Εγώ πληρώνω πολύ περισσότερα για να ταξιδέψω στην πατρίδα μου από ό,τι πριν από 5-6 χρόνια. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο βάθος του μυαλού μας. Επίσης κάτι άλλο τα άτομα μειωμένη κινητικότητας και τα άτομα με ειδικέ ανάγκες πρέπει πάντοτε να χαίρουν ιδιαίτερη προστασία και μεταχείρισης και δεν νομίζω ότι κανείς έχει αντίρρηση γι' αυτό. Με αυτά τα πέντε σχόλια λοιπόν θα ήθελα να κλείσω τα σχόλιά μου και ελπίζω ότι θα βελτιωθεί το, το, το, κείμενο. Ο πρόεδρος φοβάται ότι θα έχουμε περισσότερα παραθυράκια και κενά από ό,τι πριν. Ελπίζω πως όχι για τον κατάλογο των έκτακτων συνθήκων μπορεί να συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι εξαντλητικός ο κατάλογος, αλλά τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να το σκεφτούμε. Είναι καλό να έχουμε έναν εξαντλητικό κατάλογο του τι συνιστά έκτακτη περίσταση. Πρόεδρος, προσπαθώ να μην καταχραστώ τις θέσεις μου ως προεδρεύοντος, οπότε θα δώσω το λόγο ευθύς αμέσως στον κύριο Μπαχ. Yes, ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο για τις δηλώσεις τους και για τις εμπειρίες που μας έχουν μεταφέρει, για τις ε, συνεισφορές που έχουν φέρει και γραπτά και εδώ στην αίθουσα και θέλω να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε την άποψη της Κομισιόν και να καταλάβουμε την αιτιολόγηση των προτάσεων της Κομισιόν σε γενικές γραμμές <clears throat> νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δικαιώματα αλλά δεν είναι σαφώς καθορισμένα υπάρχει ασάφεια σε σχέση με τα δικαιώματα αυτά και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει όλους σύμφωνους ότι χρειάζεται βελτίωση της ε, σαφήνειας πολλοί συνάδελφοι θέλουν να βελτιωθεί και η νομική θέση του επιβάτη και εγώ πιστεύω κάτι τέτοιο. Προσωπικά, εγώ θέλω να εξασφαλίσω ότι οι τωρινοί κανόνες οι οποίοι υπάρχουν να ενισχυθούν με την καλύτερη διευκρίνηση. Και νομίζω ότι και η Κομισιόν χρειάζεται να, να ενισχυθεί η θέση Κομισιόν, γιατί παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι εξισορροπημένη η στάση της, εγώ θεωρώ ότι κλείνουν πιο πολύ από την πλευρά των εταιριών. Για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή μας, το είπαν και οι περισσότεροι συνάδελφοι, <clears throat> ότι θέλουμε να έχουμε ένα σαφή κανόνα, ο οποίος θα είναι απερίφραστος και να αφήσουμε μονάχα ελάχιστες περιπτώσεις αν χρειάζεται για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις. Για τις πτήσεις με ανταπόκριση. Η Κομισιόν έχει κάνει την πρότασή της σε σχέση με το χρόνο άφηξης. Τις καθυστερήσεις για το χρόνο άφηξης. Αυτό όμως σημαίνει πολλά προβλήματα για τις μικρές εταιρείες, τις περιφερειακές ε, εταιρείες, οι οποίες φέρνουν στα μεγάλα αεροδρόμια τους ε, επιβάτες και γι' αυτό νομίζω ότι τα πρώτα 90 <clears throat> λεπτά να μην υπολογίζονται για τις εταιρείε που φέρνουν στα μεγάλα αεροδρόμια. Και δεν συμφωνώ με την Κομισιόν η οποία βασίζεται μόνο σε αυτό το σημείο. Για την τιμή των εισιτηρίων είπαν ορισμένοι συνάδελφοι ότι κάπως θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια αναλογικότητα για τα φθηνά εισιτήρια να μην υπάρχει πλήρη πλήρης αποζημίωση. Εγώ θέλω να αναφέρω ότι αυτή ήταν και η θέση του Κοινοβουλίου ότι αντίθετα με τη σύμβαση του Μοντρεάλ όπου ήταν η αποζημίωση ήταν κατά και αφορούσε το γεγονός και τη βλάβη προς τον επιβάτη, προς τον επιβάτη. <clears throat> και αυτή ήταν η θέση της Κομισιόν. Εγώ είχα ζητήσει να υπάρξει μια απλοποίηση τα σημεία αυτά, τα τρία κατόφλια, 5, 9 και 12. Νομίζω ότι αυτά <clears throat> επιδεινώνουν την τωρινή κατάσταση. Εγώ προσπάθησα να εξασφαλίσω μια ορθολογικοποίηση και απλοποίηση. Το 3 και 5 νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό όπως είναι σήμερα οργανωμένες οι αεροπορικές πτήσεις. Είναι εφικτό κατά την άποψή μου. Και η απλοποίηση στα 300 και 600 ευρώ νομίζω ότι θα ήταν θετική και για τους επιβάτες. Να μπορούν οι επιβάτες λοιπόν να έχουν μια πιο απλή πληροφόρηση και επίσης <clears throat> είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της κράτησης πτήσης να αναφέρονται όλα τα στοιχεία του κόστους. Και δεν νομίζω ότι εδώ έχουμε κάποια διαφορετική άποψη. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές ε, λύσεις δεν συμμεριζόμαι τους φόβους του Πρόεδρου μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλές συμβαστικές λύσεις για να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των επιβατών χωρίς να φέρουμε <clears throat> σε μια αφόρητη θέση τις επιχειρήσεις αεροπορικές οι οποίες θα υφίστανται ένα μεγάλο άκτος. Δεν μιλάμε τώρα για τεράστια ποσά και τεράστιο αριθμό επιβατών. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό των επιβατών που είναι θύματα καθυστερήσεων και έναντι αεροπορικών εταιριών που δεν έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει <clears throat> να εξασφαλίσουμε ότι δεν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ε, ευρωπαϊκές εταιρείες εναντί των ξένων εταιριών και είμαι ε, ευγνώμων για τη συνεργασία των σχεδόν εισηγητών. Νομίζω μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Μπαχ. Κλείνει και αυτή η συζήτηση και όπως είπα και από την αρχή ο σκοπός μας είναι να ψηφίσουμε στις 17 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Το επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης είναι η χρήση εμπορικών σημάτων περιφερειακού χαρακτήρα. Είναι μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Γεωργίας από τον κύριο Ρούμπιξ. Ο κύριος Ρούμπιξ όμως δεν είναι παρόν. Ούτε κανείς άλλος από την πολιτική του ομάδα. Οπότε κάνω εγώ μια παρουσίαση ως πρόεδρος εξωρώματος του κύριου Ρούμπιξ. Μπορούμε να έχουμε λίγη ησυχία στην αίθουσα, μήπως. Ευχαριστώ. 36 τροπολογίες έχουν κατατεθεί στο σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Ρούμπιξ. Στη γνωμοδότησή μας αυτή προς την Επιτροπή Γεωργίας. Ο εισηγητής ευχαριστεί όλους αυτούς οι οποίοι έχουν καταθέσει τροπολογίες και ευχαριστεί και τους κοιόδης εισηγητές για την ε, συνεισφορά τους. Στις 24 Οκτωβρίου οι Σκιώδης συμφώνησαν σε πέντε συμβασικές τροπολογίες. Η γνωμοδότηση και οι τροπολογίες τόνισουν τον ιδιαίτερο ρόλο πρέπει να παίξει ο τουρισμός για την ανάπτυξη των σημάτων αυτών περιφερειακού χαρακτήρα, σημάτων ποιότητος. Ο εισηγητής επιμένει ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το branding αυτό, για την προώθηση των σημάτων ποιότητα θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνεργασία των κρατών μελών, ιδίω με την μεταλαμβάνευση βελτίστων πρακτικών. Οι τροπολογίε ε, <clears throat> επαυξάνουν αυτά τα οποία προτείνει ο εισηγητή και κατά την άποψη του εισηγητή μπορούν να ενισχύσουν περισσότερο τα δίκτυα εταιρική σχέση σε περιφερειακό επίπεδο. Υποστηρίζει επίση το ότι ότι οποιοδήποτε σήμα που έχει να κάνει με γεωγραφική θέση θα πρέπει να βασιστεί στα ήδη υπάρχοντα σήματα ποιότητος, της ονομασίας προέλευσης και τα διάφορα αυτά συστήματα. Δεν θέλει να υπάρξει μια νέα πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά ο Συγητή. Θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό δεν θα επιληθεί το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουν ορισμένε περιοχέ, οι οποίε είναι απομονωμένε, ή βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Μόλον τούτο, ο εισηγητή έχει προσπαθήσει να δεχτεί ως το δυνατόν περισσότερες τροπολογίε τι συμβιβαστικέ τροπολογίες που έχει καταθέσει και οι οποίε έχουν υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων. Κύριε Νταντέν, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση, όπως μας έχει υποβληθεί από τον εισηγητή μας, μας φαίνεται κάπως ασαφής, διότι το περιφερειακό σήμα ποιότητας θα πρέπει να είναι κάτι πολύ σαφώς ορισμένο. Το να έχει κανεί σήμα από τις δημόσιες αρχές θα πρέπει να σημαίνει για τον καταναλωτή ότι υπάρχει κάποια επιπλέον αξία. Και αυτό ουσιαστικά εννοούμε με την ποιότητα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρήσαμε ότι αυτή η επιδίωξη της ποιότητας θα πρέπει να είναι κάτι που να δηλώνεται σαφώς, χωρίς να υπάρχει σύγχυση και να και εμπλοκή με άλλα προβλήματα επισήμανσης. Το σήμα που μελετά αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακόμη ένα σχέδιο θεωρητικό. Αλλά θα πρέπει να βρούμε γι' αυτό το κατάλληλο, το ευστοχότερο πεδίο. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε από τον εισηγητή να λάβει υπόψη κάποιες δικές μας προτάσεις για αλλαγές, κάποιες τροπολογίες δηλαδή και πραγματικά τον ευχαριστώ που έδωσε συνέχεια στις αιτήσει και της ομάδας μας και των σκιωδών εισηγητών. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Πρόεδρος, η κυρία Μάισνερ. Äh, Ωραία είναι αυτά που είπε ο κύριος Νταντέν και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κάναμε αυτή τη συνάντηση των σχεδίων εισηγητών που ήταν πολύ θετική και εγώ συμφωνώ με αυτά που υπάρχει στην έκθεση και νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε τις τροπολογίες αυτές που ανέφερε ο κύριος Νταντέν και επίσης και με τις συμβαστικές είμαστε έτοιμοι να τις υποστηρίξουμε και μπορούμε έτσι να κινηθούμε και στην ψηφοφορία που θα γίνει αύριο. Ευχαριστώ, δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Κανείς από την Κομισιό δεν θέλει να λάβει το λόγο. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο για αυτή την έκθεση. Και τώρα έχουμε την ε, παρουσίαση από την Κομισιόν για τις νέες ε, προτάσεις στα πλαίσια των TNT. Ο κύριος Ονίλ τώρα, αν μπορούμε να τον βρούμε, θα κάνουμε την παρουσίαση. Μια στιγμή να τον βρούμε πρώτα. Πρόσκληση υποβολή εισφορών για το νέο ΔΕΔΜΗ. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ονίλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. να συνεχίσουμε αυτή την καλή συνήθεια, να ερχόμαστε και να σα ενημερώνουμε εκ των προτέρων όταν μια πρόταση βρίσκεται στο στάδιο τη ε, εκπονησή τη. Ε, ενημερώσαμε του εκπροσώπου των κρατών μελών. Μάλλον θα του ενημερώσουμε αργότερα αυτή την εβδομάδα. Τώρα μιλάμε για την τελευταία πρόσκληση στο ισχύον ε, πρόγραμμα για τα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα. Έχουμε περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα τα 70 από το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και τα 280 από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει εδώ να δοθεί έμφαση κατά πρώτον στο ποιο θα μπορέσει να μας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα, κάτι που το γνωρίζετε, δηλαδή η RTMS είναι το ένα στοιχείο και τα διάφορα προγράμματα που βελτιώνουν τις θαλάσσιες διασυνδέσεις και έπειτα η αρχή του τι δεν μας έχει δώσει επαρκή αποτελέσματα και πού θα μπορούσαν να επιτευχθούν βελτιώσεις βάσει αρκετών πρωτοβουλειών ή προγραμμάτων που ήδη μας έχουν υποβληθεί. Αυτά αφορούν περίπου το σύστημα ευθειών μεταφορών, ο φτωχός συγγενής της προηγούμενης πρόσκλησης και οι διάφορες πτυχές που έχουν να κάνουν με την καινοτομία. Σε αυτήν μας την προσπάθεια πιστεύουμε ότι έχουμε δημιουργήσει το κατάλληλο τοπίο για να καταρτιστεί η επόμενη περίοδος προγραμματισμού, η περίοδος, μάλλον το, ε, η διευκόλυνση διασυνήθως στην Ευρώπη και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να δημοσιεύσουμε αυτή την πρόσκληση ήδη από το Δεκέμβριο προκειμένου να αξιολογήσουμε και να προγραμματίσουμε εγκαίρως πριν το καλοκαίρι ποιοι θα επιλεγούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις? Τώρα είναι η ώρα να πείτε στους ενδιαφερόμενους, στους δικούς σας, να υποβάλουν τις εισφορές τους για το Δεκέμβριο. Ευχαριστούμε κύριε Νίλη. Φτάνουμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης για σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ακολούθησαν τις ε, προσκλήσεις μου για περί και μόλις συγκεντρωθούν όλοι οι συγκητές θα αρχίσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. So Δεκάλεπτο διάλειμμα για να απλώσετε τα πόδια σας, όπως λένε οι Αμερικανοί.